Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την απογευματινή μας συνεδρίαση. Ξεκινάμε λοιπόν. Καλώς σας απόγευμα. Κάποιες ανακοινώσεις θα ήθελα να κάνω, αλλά πρώτα βεβαίως πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Μερικές ανακοινώσεις λοιπόν. Υπάρχει διερμηνία διαθέσιμη σε 22 γλώσσες. Η συνεδρίαση παρακολουθείται και διαδικτυακά και σε ό,τι αφορά τα διορθωτικά για τα τεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά τεχνολογικά προϊόντα, το δεύτερο πακέτο σχεδίων διορθώσεων ε, σχετικού κανονισμού για τα in vitro και για διατροτεχνολογικά έχουν ε, φτάσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι και υπεύθυνη η Επιτροπή. Τα διορθωτικά αυτά είναι διαθέσιμα στα μέλη σε όλες τις γλώσσες και τα διορθωτικά θεωρείται ότι εγκρίνονται εκτός εάν με ως σήμερα το απόγευμα υπάρξει κάποιο αίτημα από κάποια πολιτική ομάδα, από τέσσερα τουλάχιστον μέλη, για να τεθεί προς ψηφοφορία. Έχει υπάρξει τέτοιο αίτημα από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η ψηφοφορία λοιπόν θα λάβει χώρα αύριο και για τα δύο αυτά διορθωτικά. Στη συνέχεια θα πάνε ε, προ τελική έγκριση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και θα εγκριθούν βεβαίως ε, ε, εφόσον γίνουν και οι όποιε τροποποιήσεις. Λοιπόν, θα λάβει χώρα και μια έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής ΕΝΒΗ την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Εκεί θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων πρώτα σε ό,τι αφορά την έκθεση Ευρωπαϊκό Περιβάλλον ποια είναι η κατάσταση ενώπιση του 2020 με τον εκκληστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και θα γίνει και μια παρουσίαση της ανακοίνωσης για το Green Deal, το Ευρωπαϊκό Green Deal από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Τίμερμανς. είναι σχεδόν 100% βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό ε, εφόσον όντως στις 11 Δεκεμβρίου παρουσιαστεί το Green Deal στις 16 του μήνα ο κύριος Τίμερμανς ε, θα έρθει στην Επιτροπή μας οπότε παρακαλώ να είστε εδώ ε, εκείνο το βράδυ για αυτή την πρώτη αλλαγή απόψεων. Να θυμίσω ότι έχουμε ε, και ακροάσεις σε ό,τι αφορά ε, την κοινή γεωργική πολιτική μεταρρύθμισή τη, καθώ και την, ε, τον πληθυσμό των λύκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3,5 με 6,5 με την Επιτροπή ε, Γεωργίας από κοινού για την ε, ε, μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής στο κτίριο 6Q2 και την 5η 10.30 με μία μαζί με την Επιτροπή ΠΕΤΗ, ε, αναφορών δηλαδή, για το θέμα του πληθυσμού των λύκων στο έγγραφο, στο, στην αίθουσα 3C50, συγγνώμη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Πέτερ Λίζε για ένα θλιβερό γεγονό που θέλει να μα μιλήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι συναδελφοί θα το έχουν μάθει δυστυχώ. Είχαμε μια τραγική απώλεια το, περασμένο, το προπερασμένο Σαββατοκυριακό. Ο πρώην συναδελφός Φραντσες Κάμπος ο οποίο υπήρξε για χρόνια μέλο εδώ τη Επιτροπής, ε, με μεγάλη επιμέλεια, ε, με πολύ σκληρή δουλειά, πολύ συμπαθή συνάδελφο. και δυστυχώς ε, έχασε τη ζωή του το προπερασμένο Σαββατοκυριακό και είμαι ευγνώμων. Θα ήθελα να το αποτίσουμε φορό με ένα λεπτό Thank you. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Οι ανακοινώσει του Προέδρου όσον αφορά τις συστάσεις των συντονιστών ήδη έχει κυκλοφορήσει και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης να σα κάνω μια ενημέρωση για τις τρέχουσες διοργανικέ διαπραγματεύσεις στους τριλόγους. Θα ξεκινήσω με τον τρίλογο για την ταξονομία. Μετά από την τελευταία συνεδρίαση τη Επιτροπής ΕΝΒΗ έλαβαν χώρα τρει τρίλογοι 6 Νοεμβρίου, 20 και 27 επίσης Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Η τελευταία εγώ προέδρευσα στους τρελόγους, οπότε όλα τα σημεία της δεν θα έχουν καλυφθεί. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά καλύψαμε το επίδιο εφαρμογή του κανονισμού, τους ορισμούς, τα κριτήρια για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, τη χρήση των κριτηρίων, τη διακυβέρνηση, τη κριτήρια τεχνικής, τεχνικού ελέγχου, τη ρήτρα αναθεώρησης και το καθεξής. Ο πιθανός τελικός τρίλογος θα λάβει η χώρα αύριο. τον οποίο θα συμπροεδρεύουν οι ΕΝΒ και οι ΕΚΟΝ. Επίσης έχουμε τριλόγους για την ποιότητα των υδάτων και τις ελάχιστες απαιτήσει για την επαναχρήση νερού. Όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού, ο τρίτος τρίλογος έλαβε χώρα στις 19 Νοεμβρίου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημείωσαν αργή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Συμφώνησαν προσωρινά μόνο για το κομμάτι που αφορά την προσέγγιση βασική επικινδυνότητας. Προχώρησαν συζητήσεις για την πληροφορία σε πληροφορίε, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό, την πρόσβαση στα ύδατα και συγκεκριμένε παραμέτρου ειδικότερα το μόλιβδο τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα μικροπλαστικά. Πολλά πολιτικά θέματα όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, τα μικροπλαστικά, ε, ο μόλιβδος, ε, η καταξιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και ούτω καθεξής πρέπει από μένα να επιληθούν. Δεν πρόκειται να αλλάξει ιδιαίτερα θέση στο Συμβούλιο, οπότε είναι αρκετά απίθανο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στον τρίλογο αυτής της εβδομάδας ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί ως τελευταίος για την ταξονομία. Ο δεύτερος τρίλογος που σχετίζεται με τα υδάτα, ελάχιστες απαιτήσει για την επανάχρηση των υδάτων. στις 12 Νοεμβρίου έλαβε χώρα ο δεύτερο τρίλογος για τι ελάχιστες απαιτήσει για την επανάχρηση νερού. Σε αυτόν τον τρίλογο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζήτησαν σε βάθο διάφορα ειδικά ζητήματα επιτεύχθη προσωρινή συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ενώ παρα, η συμφωνία για το αντικείμενο, το ευρώ και το πεδίο εφαρμογή. Περαιτέρω, συζητήσει απαιτούνται για τι υποχρεώσει όσον αφορά του φορεί ε, ε, υδάτων όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων, του ελέγχου συμμόρφωση και τα παρατήματα 1 και 2. Οι θέσει των συνομοθετών διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, τι υποχρεώσει όσον αφορά τις, ε, την επανάχρηση αδειών, οι εξουσιοδοτήσει και την πρόσβαση σε, την προσφύγη στη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να απογορέψουν οικονομικέ δραστηριότητε που εφαρμόζουν την επανάχρηση υδάτων. Απόψε το βράδυ θα γίνει ο τρίτο τρίλογο. Πάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης και καλωσορίζω τον κύριο Χάνσεν, τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΚΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Είναι η ετήσια επίσκεψή σας. Ε, αν και είχατε έρθει πριν από δύο εβδομάδες, ε, δεν είναι και άσχημη η συνήθεια αυτή. Έχετε 10 λεπτά για να μας παρουσιάσετε το έργο σας, τις προτεραιότητές σας και μετά θα ανοίξουμε, θα δώσουμε το λόγο στα μέλη. Παρακαλώ. Very much, Mr. Chairman, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ακροατήριου. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά εδώ μετά από δύο εβδομάδες μαζί με όλους τους οργανισμούς ε, που αναφέρονται εδώ στην Επιτροπή. Σας έχουμε συστηθεί και αυτή τη φορά είμαι μόνος μου. Στον ετήσιο μας διάλογο, όπως ονομάζεται, για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του έργου της ΕΚΑ το τελευταίο έτος και να ρίξουμε και μια ματιά προς το μέλλον. Στην τελευταία μας συζήτηση πριν από ένα χρόνο, το βασικό μήνυμα που αποκόμισα εγώ ήταν ότι η Επιτροπή αυτή φυσικά σε ένα διαφορετικό σχηματισμό είχε σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτό που ονομάζουμε ελέγχου ε, συμμόρφωση. Κάτι που διαβάζουμε συχνά στον τύπο με αφορμή κάποιε μελέτες ε, που έχουν γίνει που βασίζονται σε διάφορα δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί στο ΡΙΤΣ και λέγεται ότι αυτά τα δεδομένα δεν, είναι, ε, δεν συμμορφούνται με τις απαιτήσει. Και εγώ υποσχέθηκα ότι θα εντείνουμε τις εργασίες μας όσον αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης και τότε δεν ήθελα να σας δώσω έναν αριθμητικό στόχο αλλά ελπίζω να μπορέσω να σας δώσω τις σχετικές πληροφορίες ικανοποιητικά σήμερα. Το άλλο που συνέβη ε, σε σχέση με την Επιτροπή σας το τελευταίο έτος αφορά την εξουσιοδότηση του ΡΙΤΣ όπου υπήρξε πάλι ένα ψήφισμα ως αντίρρηση απόφασης της Επιτροπής ε, που έδινε απόφαση στις εξουσιοδοτήσεις και όσον αφορά αυτό το ψήφισμα έγιναν κάποια σχόλια για τη δουλειά που κάνουμε στην ΕΚΑ. Το ψήφισμα αυτό από τη δική μας άποψη και όσον αφορά τα θέματα που τέθηκαν αποτελούσε συνέχιση πολλών άλλων διαφορετικών ψηφισμάτων που έχουν προέρθει από αυτό το Κοινοβούλιο και που συνάδει απόλυτα με την απόφαση του δικαστηρίου που εκδόθηκε την Άνοιξη και που επικρίνει ακριβώς τους ίδιους ε, παράγοντες. Οπότε θα σας αναφέρω και για αυτό, για το τι έχουμε κάνει. Ας ε, πάμε όμως πίσω στη στρατηγική. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο υιοθέτησε στα τέλη του 2018, δηλαδή λίγο μετά από τον τελευταίο μας διάλογο, ένα στρατηγικό σχέδιο για τα έτη 2019 έως 2023. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τρεις στρατηγικές προτεραιότητες. Ε, ε, για να σας τη συνοψίσω, η πρώτη είναι προσδιορισμός ανησυχητικών ουσιών και ανάληψη δράσης γρήγορα. Το δεύτερο στρατηγικό σχέδιο είναι η υποστήριξη της βιομηχανίας στην απόκτηση πληροφοριών που έχουμε εμείς στην ΕΚΑ και που έχουν οι ενδιαφερόμενοι στις εταιρείε σε όλη την αλυσίδα παραγωγή, ότι σε αυτό που χρησιμοποιεί πραγματικά την ουσία να έχει στη διάθεσή του τις που χρειάζεται για να προστατεύσει αυτό εαυτό του και για του καταναλωτέ όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντο. Και ο τρίτη, η τρίτη στρατηγική προτεραιότητα είναι εμεί ω οργανισμό να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά που κάνουμε ε, ενσωματώνεται καλύτερα στο ευρύτερο πλαίσιο των άλλων νομοθετημάτων ε, που εφαρμοζούνται από άλλους ε, και στη διεθνή ατζέντα. Τι έχουμε επιτύχει λοιπόν. Αν δούμε τις τρεις στρατηγικές προτεραιότητες, θα αναφερθώ πρώτα στην πρώτη. Έχουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την αλυσίδα προμηθειών και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στη δύο ε, θα σας αναφέρω ότι έχουμε επιτύχει επίση και στην τρίτη τρία κάποια από που έχουμε καταφέρει διότι στις κατευθυντήριες γραμμές ε, τη Πρόεδρου Ursula von der και ειδικότερα στο πλαίσιο του Green Deal και τη ατζέντα για μηδενική ρήπανση, διακρίνω διάφορε δυνατότητες που έχουμε εμεί στον οργανισμό μας να υποστηρίξουμε το έργο τη επιτροπή. Ξεκινώντας από τη συμμόρφωση, ο στόχος ο οποίος είχαμε εμείς ε, πέρυσι για το 2018 ήταν 2.200 ε, έλεγχοι συμμόρφωσης ε, και με χαρά μου μπορώ να σας πω ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στους 300 ή πάνω από 300 φέτος. Έχουμε αυξήσει λοιπόν τον αριθμό των ελέγχων σε πάνω από 50%. Έχουμε ολοκληρώσει 283 ε, συγγνώμη, 200 ελέγχους εμόρφωσης για 283 ουσίες ε, για 218 άδειες. Ε, ε, έχουμε μεγάλη αύξηση λοιπόν σε σχέση με πέρυσι και ελπίζουμε ότι αυτό να σας ικανοποιεί ως σημαντική αύξηση όπως σας είχα υποσχεθεί στην Επιτροπή σας πέρυσι. Όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις, έχουμε κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συντάσσουμε τις γνωμοδοτήσεις και τις πληροφορίες που δίνουμε εμείς στην Κομισιόν ώστε να ε, ευθυγραμμιζόμαστε με τα δικά ψηφίσματα, αλλά και με την αποφάση του δικαστηρίου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, εκτός αν μου κάνετε ερωτήσεις. Απλά έχουμε ευθυγραμμιστεί με αυτό που μας ζητήθηκε, ώστε να σεβόμαστε και τις απόψεις που εκφράσετε εσείς και ε, τις απόψεις του δικαστηρίου. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι εμείς τα κάναμε όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα έχουμε τεράστιο αριθμό αιτήσεων για εξουσιοδοτήσεις. 120 τρέχουν αυτή τη στιγμή προς διεκπαιρέωση ε, στο δικό μας σύστημα. Αυτό συγκριτικά με τους 22 που είχαμε την τελευταία φορά που ήμουν εδώ το 2018. Οπότε έχουμε 500% αύξηση, πενταπλάσια αύξηση των αιτήσεων για εξουσιοδοτήσεις. Χρειάστηκε λοιπόν να επιταχύνουμε σημαντικά, να αυξήσουμε τον αριθμό του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα αυτό και να αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Όσον αφορά του περιορισμού, έχουμε συνεχίσει ε, τι εργασίε μα πολύ εντατικά. Έχουμε πολλέ προτάσει περιορισμών που βρίσκονται υπό διεκπαιρέωση τώρα ε, θα σας πω κάποια ονόματα, κάποιους αριθμούς. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τέσσερις στην ΕΚΑ. Αφού μας το ζήτησε ε, η Κομισιάν, έχουμε εννέα περιορισμούς που συζητώνται αυτή τη στιγμή στις διάφορες επιτροπές και έχουμε και πέντε προτάσεις περιορισμών που έχουμε στείλει στην Κομισιόν και που ε, έχουν μπει σε διαδικασία λήψη απόφαση και για να σας αναφέρω κάποια σημεία αφορά τη μελάνη για τα τουάζ, ε, ένα τομέα που δεν έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει, ε, ρυθμίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια χημικά επιτρέπονται και ποια όχι, για τη μελάνη για ε, τα έχουμε μια άλλη για τα μικροπλαστικά που τρέχει αυτή τη στιγμή και άλλη μια για τα για ελαστικά που χρησιμοποιούνται ε, στο τέλος της ζωής των ελαστικών σε γήπεδα αγώνων σε αθλητικούς χώρους. Ε, όπως σας είπα, είναι, εργαζόμαστε με μεγάλη ένταση και βάσει αυτών των εργασιών και γνωρίζοντας ε, τι εργασία θα πρέπει να κάνουμε, αυτό που κάναμε στον οργανισμό μας είναι ότι αναδιοργανωθήκαμε σημαντικά, ούτω ώστε να προσαρμοστούμε στις προκλήσεις αυτές, τόσο σε αυτές που αφορούν τους ελέγχους συμμορφώσεις, ε, τους περιορισμούς και τις οξυσοδοτήσεις, αλλά και με στόχο να προσπαθήσουμε να βρεθούμε σε μια καλύτερη θέση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νέα καθήκοντα. Ο οργανισμός μας δηλαδή ως οργανισμός, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε ε, οργανώνεται βάσει τριών αξώνων. Ο ένας αφορά κέντρα ε, ικανοτήτων, ο δεύτερος είναι ότι ολόκληρος ο οργανισμός έχει ε, οργανωθεί έτσι ώστε να αρχίσει να ερευνά ομάδες ουσιών, δηλαδή τακτικά εξετάζει πολλές ουσίες μαζί και όχι μεμονωμένα και τέλος, με αυτή την οργάνωση σε ομάδες ουσιών και ικανοτήτων πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να αναλάβουμε νέα καθήκοντα πολύ πιο εύκολα. Τι σημαίνει αυτό το ευκολότερα, ότι μπορούμε να ξεκινάμε ταχύτερα, με λιγότερες δυσκολίες από ό,τι παλιότερα. Από τα νέα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει, να σας αναφέρω κάποια, Τώρα με τα κέντρα δηλητηρίων έχουμε ξεκινήσει. Μιλάμε για βάση δεδομένων και συλλογή δεδομένων από βιομηχανία, όπου ξαναδίνουμε τις προφορές αυτές στα κράτη-μέλη, ώστε ε, οι αρχές αντιμετώπισης ε, έκτακτης ανάγκης μέσω τηλεφώνου να μπορούν να συμβουλέψουν ε, τον κόσμο για τη χρήση χημικών σε περίπτωση δηλητηρίασης. Επίσης προχωράμε πολύ καλά στο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη βάση δεδομένων ε, για τα απόβλητα που συζητήσαμε την περασμένη φορά ως μια κρίσιμη βάση δεδομένων ότι πρέπει οπωσδήποτε να ε, ολοκληρωθεί και να αρχίσει να τρέχει, η πρόοδος είναι ικανοποιητική. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε πλέον να αναλαμβάνουμε ε, καθήκοντα που μας στέλνει η DG Employment για την έκθεση στον εργασιακό χώρο και τις σχετικές τιμές. Όσον αφορά τη στρατηγική προτεραιότητα 2, να σας αναφέρω τι κάνουμε εκεί στην αλυσίδα προμηθειών Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες ε, για να λαμβάνουμε αποτελεσματικά πληροφορίες από τις χιλιάδες εγγεγραμμένους. Ε, πάρα πολλές πληροφορίες για χημικά. Ε, προσπαθούμε η συλλογή αυτή να γίνεται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά και να φτάνουμε μέχρι τις εταιρείε που χρησιμοποιούν τα χημικά. Οπότε έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο σε επίπεδα REACH. Τώρα βρισκόμαστε σε συνομιλίε με τα κράτη-μέλη και με την Κομισιόν γιατί ένα από τα μεγάλα εμπόδια που παρεμπόδιζε τη χρήση αυτών των πολύτιμων πληροφοριών από τους εργαζομένους ε, που εργάζονται με αυτές τις ουσίες ήταν η επαφή με την νομοθεσία ε, εργασιακών ε, κινδύνων για την υγεία. Οπότε πρέπει να άρουμε αυτά τα εμπόδια για να μπορέσουμε να ε, ε, έχουμε σε αποτέλεσμα όλα τα ωφέλη για τους εργαζομένους από αυτές τις πληροφορίες που δημιουργούνται από το REACH. Τέλος, αυτό που θα μπορούσα να σας πω για τη στρατηγική προτεραιότητα 3, που αναφέρεται στη σχέση με άλλου ε, νομοθετήματα αλλά και με το τι συμβαίνει διεθνώ, ε, ένα βασικό βήμα που επιτύχαμε ήταν η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια των Τροφίμων. Υποστηρίζουμε τον ΕΦΣΑ για την υλοποίηση τη νέα νομοθεσία για τα τρόφιμα, ειδικότερα μέσω τη υποστήριξη και ανάπτυξης συστηματοπληροφορικής συλλογή και δημοσίευση δεδομένων στο διαδίκτυο, όπω απαιτείται από την νομοθεσία για τα τρόφιμα. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια πολύ απτή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Θα χτίσουμε ίδια συστήματα, ταυτόσιμα συστήματα για την ΕΚΑ και την ΕΦΣΑ για τους σκοπούς αυτούς και έτσι θα χρησιμοποιήσουμε και συνέργειες αλλά και θα κάνουμε τη δουλειά μας με μεγαλύτερη συνοχή. Τώρα κοιτώντα προς το μέλλον, τι πρόκειται να γίνει στην επόμενη διετία, σαφώς για την ΕΚΑ έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και όπως είπα, οι έλεγχοι συμμόρφωσης που κάνουμε έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και σκοπεύουμε να τους διατηρήσουμε έτσι για την επόμενη επταετία. Ούτω ώστε να μπορούμε να πούμε το 2027 ότι έχουμε εξετάσει όλες τις ουσίε ε, που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουμε καθορίσει κατά πόσο χρειάζεται διαχείριση κινδύνου ή όχι για την καθεουσία. Παρατηρούμε ότι ε, στο πλαίσιο τη Πράσινη Συμφωνία αυτό που εμείς καταλάβουμε από αυτή τη συμφωνία είναι ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία να απλουστεύσουμε την νομοθεσία για τα χημικά μαζί με τις συστάσεις που υπάρχουν στους ελέγχους καταλληλότητας όλης της, ε, της Κομισιόν για όλες τις ουσίες ε, συμπεριλαμβανομένου του ΡΙΤΣ με αποτέλεσμα πιο αποτελεσματική δουλειά και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων που αφορούν τα χημικά, μειώνοντας έτσι τον ε, φόρτο για τις επιχειρήσεις, αλλά και αυξάνοντας την προστασία. Τέλος, μία σημείωση για τους πόρους. Μας ανησυχούν ε, οι τυχόν περικοπές που μπορεί να επέλθουν δεδομένου ότι η ζήτηση όπως φαίνεται θα παραμείνει όπως έχει σήμερα. Και είμαι βέβαιο, ε, όπω έχω ακούσει από εσά σήμερα, θέλετε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά στο πλαίσιο τη συμμόρφωση, πολλή δουλειά στο πλαίσιο των εξοδοτήσεων, πολλή δουλειά στο πλαίσιο των περιορισμών και θέλετε να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε θα προκύψει ω εξέλιξη πολιτικά για τον Green Deal και την ε, ατζέντα για τη μηδενική μόλυνση. Οπότε, δεδομένων αυτών, ε, προσδοκώ ότι θα χρειαστούμε κάποιο είδου σταθερή παροχή πόρων στην ΕΚΑ, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πρόταση της Κομισιόν. Αν θέλετε να συζητήσουμε οποιασδήποτε λεπτομέρειε, ευχαρίστω να τι συζητήσουμε στη συνέχεια. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω την εισαγωγή μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ε, ο υπεύθυνο επικοινωνία ε, με την υπηρεσία σα, ο Μάρτιν Χότζικ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην Πράσινη Συμφωνία και αναρωτιέμαι ποια είναι η εμπλοκή από την πλευρά της Επιτροπής. Και ελπίζω ότι ήδη η Επιτροπή σκέφτεται πώς θα γίνει αυτό. Θα ήθελα όμως να ακούσω και περισσότερα πράγματα από εσά για το πώς βλέπετε τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας σε σχέση με την καινοτομία που μπορεί να επέλθει ώστε να έχουμε πιο ασφαλή χημικά προϊόντα αλλά και τα θέματα της ασφάλειας των καταναλωτών ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εισαγωγής προϊόντων από την Κίνα και την όλο και αυξανόμενη διαδικτυακή αγορά. Ποια είναι η άποψή σας, πώς μπορεί η ΕΚΑ να βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση πρώτα. Ε, ως ε, σημείο επαφής έχετε εσείς αυτό το πλεονέκτημα και συνέχεια θα ακολουθήσουν οι άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάρτιν. Θα ξεκινήσω γενικά με την Πράσινη Συμφωνία. Η δική μας η εμπλοκή έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή και στη συνέχεια η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις. Η βασική μας γραμμή βασίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην κυκλική οικονομία και δεύτερον, στην καλύτερη ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι, υπάρχουν περίπου 40 νομοθετικά εργαλεία, κείμενα, που έχουν να κάνουν με τα χημικά προϊόντα και εν γέννη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ε, με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές επί συγκεκριμένων προϊόντων. Θεωρώ λοιπόν ότι αναλύοντας αυτή την νομοθεσία και φέρνοντάς το αυτό στην Επιτροπή, θεωρώ ότι μπορούμε να ε, λάβουμε ε, καλύτερα υπόψη μας ε, άλλη νομοθεσία. Για παράδειγμα, υπάρχει η οδηγία για τα ύδατα που θέτει κάποια, κάποια πρότυπα για την ε, ποιότητα των υδάτων. Υπάρχει ο περιορισμός των επικίνδυνων χημικών ουσιών στα απόβλητα, για παράδειγμα. Και το θέμα του πόσιμου νερού και η νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τριμερής διάλογος στον οποίο μπορούμε να εμπλακούμε. Όλα αυτά λοιπόν τα νομοθετικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και στόχος είναι να τα υποστηρίξουμε ώστε να, δημιουργούν, να δημιουργηθούν συγγνώμη, συνεργασίες. Και συνεργασίες μας βοηθούν να μην δίνουμε αντικρουόμενα μηνύματα. Ένα χημικό προϊόν ε, είναι ένα χημικό προϊόν ανεξάρτητα με το πώς χρησιμοποιείται. Σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, εγώ θεωρώ ότι η κυκλική οικονομία έχει να κάνει με την κυκλική χρήση των υλικών και τα υλικά είναι μία μίξη χημικών προϊόντων. Η διασφάλιση λοιπόν ε, της ασφάλειας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κυκλική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορούμε φυσικά μέσω της καινοτομία να έχουμε κυκλικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην ανακύκλωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προκλήσεις της καινοτομία. Σε γενικές γραμμές, η αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το REACH, ε, ο κανονισμός REACH είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ο κανονισμός ε, CLP για τα βιοκτώνα. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί έχουν ως στόχο να πάμε από τις πιο επικίνδυνες ουσίες στις λιγότερο επικίνδυνες ουσίες. Στη διαδικασία αδειοδότησης του χρωμίου, για παράδειγμα, έχουν υπάρξει κάποιες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για το χρώμιο 6 το χρώμιο 3 το οποίο δεν ενέχει τόσους πολλούς κινδύνους. Η πρακτική εφαρμογή όλων αυτών προωθεί την καινοτομία προφανώς, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα εφόσον υπάρχουν οι πόροι. Είμαστε σε καλό δρόμο για την προώθηση της καινοτομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η καινοτομία θα πρέπει να προωθηθεί σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία. Τώρα, εμείς στην ΕΚΑ αυτό που κάνουμε είναι ότι συντονίζουμε τους υπευθύνους εφαρμογής των πολιτικών και στόχος φυσικά είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προστατεύονται τα σύνορα από παράνομα προϊόντα που προέρχονται όπως αναφέρατε για παράδειγμα από την Κίνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιος θα ζητήσει το λόγο. Οποιο ενδιαφέρεται, ο Πίτερ Λίζε πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Χάντζεν. Αναφερθάτε κάποια σημεία πολύ συγκεκριμένα, ε, τα οποία θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο και να κάνω μετά μια γενική ερώτηση βάσει αυτών. Αναφέρατε το χρώμιο και εδώ στο Κοινοβούλιο τον είδαμε, το εξετάσαμε τον προπερασμένο μήνα. Είχαμε μια απόφαση με μικρή διαφορά στην ψηφοφορία. Έχω δει πως το έχει αξιολογήσει η Κομισιόν. Ε, υπάρχει, είναι αναπόφευκτη κάποια περιεκτικότητα σε χρώμια και θέλω να μου πείτε, έχετε ελέγξει τις εναλλακτικέ. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην τροπολογία που ψηφίσαμε εμείς τον Οκτώβριο. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε κάποια εναλλακτική. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν και συζητήσαμε πάρα πολύ και με τους προκατόχους για το ερώτημα του τι μπορεί να γίνει με αυτό. Να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλη αυτή την απέτηση. Μας είπαν ότι δεν υπήρχε καμία εναλλακτική Όπω φαίνεται, κανεί δεν την ξέρει αυτή την εναλλακτική, ενώ θα έπρεπε να την γνωρίσουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα ελαστικά. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της κυκλικής οικονομίας και την ανάγκη να μειωθούν ε, οι επικίνδυνες ουσίες. Εγώ ξέρω ότι από τα παλιά λάστιχα, όπως ξέρω, δεν αποτελούν κίνδυνο ε, για έκθεση ε, επικίνδυνων, ανθρώπων σε επικίνδυνα χημικά. Διότι μπορεί κανείς να βγάλει αυτές τις χημικές ουσίες μέσα στα χρόνια από την παραγωγή. Ε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν κίνδυνος για τους ανθρώπους, πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και κάποια συμβαστική λύση. Το τρίτο χαίρομαι που συνεργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, διότι οι περισσότερε ουσίε αποτελούν κίνδυνο κατά τη διάρκεια τη παραγωγή. Στι διαδικασίε παραγωγή εκεί χρειαζόμαστε πολύ αυστηρού κανόνε. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποτελεί όμω αυτό πρόβλημα για τον τελικό χρήστη. Οπότε πρέπει να βρούμε μια λύση για του κανόνε εργασία για του εργαζομένου και να ε, κάνουμε πιο αυστηρή την νομοθεσία. Thank you. You Ευχαριστώ από την S&D τώρα, η επόμενη ομιλητρία. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, ε, κύριε Διευθυντά. Έχουμε ήδη μελετήσει, εξετάσει μια μελέτη μάλλον του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση Κινδύνου και την Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος που, που, που δείχνει ότι ένα τρίτο των προϊόντων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 παραβιάζουν την κοινωτική νομοθεσία προστασίας ε, του περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπων από την έκθεση, δηλαδή την επιζήμια. Μόλις ένα μικρό ποσοστό συμμορφώνεται, ενώ τα υπόλοιπα χρήζουν ακόμα περαιτέρω εξέταση. Ο κανονισμός REACH υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αναφέρουν κατά πόσο οι ουσίες τους είναι καρκινογόνες, έχουν τοξικά στοιχεία, ε, δημιουργούν βιοσυσσόρευση, ε, κάνουν κακό στα παιδιά ή στη γονιμότητα. Ε, δεν μπορούμε να αγγιόμαστε ε, για προϊόντα όταν χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να φτάσουμε σε συμπεράσματα για τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου. Συμφωνείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, ότι η Ευρώπη δηλαδή στην Ευρώπη υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες ουσίες ή τις οποίες εμείς ε, επιτρέπουμε να κυκλοφορούν στην Ευρώπη χωρίς να υπάρχουν απαραίτητε πληροφορίες και τι θα γίνει με τη συμμόρφωση. Όταν δούμε το σχέδιο δράσης, ε, πριν το δούμε μάλλον, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για ποιες δράσεις ε, σκοπεύετε να διενεργήσετε. Επίσης, γνωρίζω ότι μόλις 20% όλων των αιτήσεων έχουν δοκιμαστεί στην Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό. Και κάτι ακόμα, δύο ακόμα ερωτήματα σημαντικά και αυτά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, για την προσέγγιση της ομαδοποίησης. Ε, θα συγκρίνετε τις νέες ουσίες ε, με χαμηλότερα μεγέθη σε σχέση με τις παλαιότερες, αν κατάλαβα καλά, εντός του επόμενου έτους. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πιο λεπτομερό σκοπεύετε να κάνετε και τέλος για τα μικροπλαστικά. Όπως γνωρίζετε η ΕΚΑ πρότεινε την απαγόρευση μικροπλαστικών σε προϊόντα όπως οδοντόπαστα, καλλιντικά κτλ. Ε, πότε θα έχουμε μια εικόνα για, το, για τις δράσεις που θα αναλάβετε προς την κατεύθυνση αυτή. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Για τους πράσινους τώρα, η Ιούτα Πάρις. Χαίρομαι που ξαναβλέπω και Χέντεν, χαίρομαι που ξαναήρθατε. Ε, για να μας ενημερώσετε για το έργο σας. Κάποια από τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω έχουν ήδη τεθεί από συναδέλφους και εγώ θα ήθελα να γνωρίζω ποιο είναι το ποσοστό των φακέλων REACH που ε, μελετώνται, εξετάζονται σήμερα. Ε, πρέπει να φτάσουμε στο 20% όπως γνωρίζουμε. Πού βρισκόμαστε όμως αυτή τη στιγμή ε, και πότε πιστεύετε εσείς ε, ότι οι φάκελοι αυτοί θα συμμορφωθούν πλήρως ε, για να μην έχουμε αυτά τα υψηλά ποσοστά στην οποία αναφέρθηκε ήδη η κυρία Γκούντελαντ. Ε, και κάτι άλλο για τις άδειες. Στην τελευταία θητεία αλλά και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες αδειοδοτήσεις που είναι προβληματικές. Το χρώμιο 6 παραδείγματο χάρη. Όταν ο ετών δεν προσκομίζει ένα πλήρη φάκελο με όλες τις ε, πληροφορίες τότε δεν πρέπει να λαμβάνει η χώρα διοδότηση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Επίσης, ε, διαπιστώνω ότι δίδονται κάποιες ε, ε άδειε ε, για λόγω οικονομικών συμφερόντων. αλλά αυτό πρέπει να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, μια αξιολόγηση σωστή των ενδεχόμενων υποκατάστατων ε, υπάρχει, γιατί εγώ δεν έχω δει. Επίσης, αντί να δίνουμε άδειες ε, ε γιατί να μην δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία για τα υποκατάστατα αυτά. Ε, και τέλος θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απόψή σας ε, για το, σύστημα, το, το ζήτημα του διοξιδίου τιτανίου που θα συζητήσουμε και αργότερα σήμερα. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ, η Άνια Άζεκαμπ. Ευχαριστώ τον κύριο Χάνσεν για την παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα καλλιντικά και το σχετικό κανονισμό έχω ένα ερώτημα. Ο σχετικό κανονισμός του 2013 ε, απαγορεύει τις δοκιμές σε ζώα για τα καλλιντικά και τα συστατικά τους. Είχε, έχει στεφθεί από επιτυχία αυτή η ψηφοφορία, αυτή, αυτός ο κανονισμός. Όμως παρόλα αυτά ξεκολουθούν να λαμβάνουν τέτοιες δοκιμές ε, και, και καλλιτικών και συστατικών καλλιντικών ε, στα πλαίσια του κανονισμού για τα χημικά και για το REACH όταν υπάρχει η δυνατότητα ε, όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεση του εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένε ουσίε, ε, συμβαίνει αυτό και ανεξάρτητα μάλιστα από την έκθεση ε, εργαζομένων σε κίνδυνο που χρησιμοποιούνται ζώα. Ε, εδώ ε, δημιουργείται κίνδυνος. Είναι σαν να λέμε στην πραγματικότητα ότι ο κανονισμός REACH υπερτερεί το κανονισμό για την απαγόρευση δοκιμών σε ζώα και χωρίς να ενημερώνεται και καταλήλως ο καταναλωτής. Συμφωνείτε κύριε Χάνσεν ότι οι πρακτικές που ακολουθείτε στα πλαίσια του κανονισμού REACH υπονομεύουν τον κανονισμό για την απαγόρευση δοκιμών πάνω σε ζώα σε ό,τι αφορά τα καλλιντικά. Ε, και τι σκοπεύετε να κάνετε αυτό, διότι και εδώ υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή. Ευχαριστούμε. Ε, πάμε πίσω στο ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Χάνσεν. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, ήταν εξαιρετική. Αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα της δουλειάς σας λαμβάνονται υπόψη. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες. Και αν ναι, ποιος εποπτεύει. Έχω κάνει αυτή την ερώτηση πολλές φορές σε διάφορα φόρα δεν έχω ωστόσο λάβει κάποια ικανοποιητική απάντηση ακόμα. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνα χημικά. Δηλαδή ποιος πραγματοποιεί την εποπτεία και οι δικές σας αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη στις εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Τελευταία από την κυρία Σπυράκη, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια περίεργη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε για το διοξείδιο του τιτανίου που συζητάμε. Ε, θέλω να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες. Πρώτον, θα ήθελα να μου πείτε ποιο χρονοδιαγράμμα προβλέπετε για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τα απόβλητα από την DGMV όσον αφορά το διοξείδιο του Διτανίου και την ε, ταξινόμησή του γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε τις κατευθυντές γραμμές ε, όταν ε, η ε, ταξινόμηση τεθεί σε ισχύ για να αποφευχθούν προβλήματα. Και όσον αφορά τις δικές σας αρμοδιότητες, ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πρώτα στο σχέδιο γίνεται αναφορά για τα υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά. Υπήρχε μάλλον αναφορά, αλλά τώρα έχει καταργηθεί. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Και δεύτερον, ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την εκθεσή σας για το διοξείδιο του τιτανίου, είστε έτοιμοι να δώσετε κάποια διευκρίνηση όσον αφορά το παράρτημα 3, σημείωση 10, όπου έχετε βάλει τη λέξη dry μπροστά από τη λέξη powder όσον αφορά και τα ποσοστά, διότι όπως αναφέραμε υπάρχουν έργα εδώ πέρα ε, όσον αφορά την ε, κατοχή ε, και την επεξεργασία τιτανίου, όπου υπάρχει διοξείδιο του τιτανίου και μπορεί να περάσει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω τη όσφρηση. Έχετε κάποιε προφορέ γι' αυτά. Πολλέ, πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει λοιπόν. Οπότε θέλουμε να δώσετε και πολύ συγκεκριμένε απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ξεκινάμε τον έλεγχο συμμόρφωσης, την αδειοδότηση Πρώτα τον έλεγχο τη μετά τι αδειοδοτήσει και μετά κάποια από τα ζητήματα που αφορούν του περιορισμού. Και μετά θα πάμε στα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, την απασχόληση, τα καλλιντικά και το διοξείδιο του τιτανίου. Όσον αφορά τους ελέγχους συμμόρφωσης, ναι, συμφωνήσαμε με την Κομισιόν ότι θα αυξήσουμε την ποσότητα των φακέλων που ελέγχουμε για θέματα συμμόρφωσης από 5% σε 20%. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση στην αρμόδια επιτροπή και η, η οποία την ενέκρινε. Οπότε έχουμε αύξηση του ποσοστού διεκπαιρέωσης από 5% σε 20%. Αυτό αφορά τον αριθμό των φακέλων. Εμείς αυτό παραμένουμε ότι αν δούμε τον αριθμό ουσιών που καλύπτει αυτό, και αν θέλετε θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο. Αντιστοιχεί σε κάπου μεταξύ 30 ε, έως 40% όλων των ουσιών που έχουν καταχωριστεί. Αυτές θα εξετάζουμε μέσω των ελέγχων συμμόρφωσης. Για όλες τις υπόλοιπες ουσίες θα τις εξετάσουμε από την εξή προοπτική κατά πόσο θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει σχετική διαχείριση ε, κινδύνου άμεσα, δηλαδή χωρί ανάγκη δημιουργία περαιτέρω δεδομένων, κατά πόσο μπορούμε να πάμε κατευθείαν δηλαδή στην κατηγοριοποίηση και την επισήμανση ε, σε περιορισμούς, με αποτέλεσμα περιορισμού ή αδειοδότηση ή κάποιο άλλο είδου εργαλείο όπω όρια έκθεση, ή αν θεωρούμε ότι έχει γίνει επαρκής έλεγχος επικινδυνότητας οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω δουλειά για την ουσία για κάποια ουσία. Και μετά υπάρχει ένας τρίτος τύπος ε, ε, συμπεράσματο ή ομάδα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που, όπου θα καταλήξουμε. Το ότι βλέπουμε μια ουσία, θεωρούμε ότι δεν είναι ανησυχητική, ωστόσο τα δεδομένα μπορεί να μην συμμορφούνται. Δεν θα μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες τώρα για ποιο είδους ουσίες ε, ανήκουν σε αυτή την περίπτωση, αλλά κάποιες ουσίες γενικότερα θεωρείται και οι εμπειρογνώμονες μας συμφωνούν, δεν είναι τοξικές, ωστόσο στο πλαίσιο της καταχώρησης ε, ε, αυτό δεν αποδεικνύεται πολύ καλά. Οπότε τέτοιου είδους ουσίες θα έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα, αλλά φυσικά θα συζητήσουμε με τους υπευθύνους καταχώρησης, ούτω ώστε να βελτιώσουν τους φακέλους καταχώρηση. Στόχο είναι μέχρι το 2027 να έχουμε εξετάσει όλε τι καταχωρισμένε ουσίες ε, οι οποίε να έχουν περάσει από ελέγχου συμμόρφωσης, από διαδικασία διαχείριση ε, κινδύνου ή να καταλήξουμε ότι δεν χρειάζεται διαχείριση κινδύνου γιατί είναι ασφαλέστατε βάσει ε, αδειάστη ή υπάρχουν άλλε ε, που, δεν είναι, που δεν συμμορφούνται αλλά που δεν χρειάζεται για τι οποίε δεν χρειάζεται να εξάγουμε δεδομένα, να γίνουν σχετικέ ε, δοκιμές, γιατί θα κόστιζε πάρα πολύ σε πόρους, σε, σε χρήση μέσων για να γίνουν σχετικέ δοκιμέ. Όπω είπα, όλα αυτά θα έχουν γίνει μέχρι το 2027. Όσον αφορά τι αδειοδοτήσει, να δούμε και την ομοδοποίηση εδώ ταυτόχρονα. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε, μάλλον το κάνουμε ήδη, αλλά θέλουμε να γίνεται πιο συστηματικά από την 1η Ιανουαρίου του 2020, θα είναι ότι όλες οι ουσίες που εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τις δικές μας διαδικασίες αξιολόγησης, περιορισμού, αδειοδότησης ε, ή που αφορούν οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα, θα εξετάζουμε όλες τις, ε, ταυτόχρονα όλες τις ουσίες που χημικά είναι παρόμοιες ακόμη και εκείνες που δεν έχουν καταχωριστεί καθόλου, για να δούμε κατά πόσο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε πιο ε, αξιόπιστα συμπεράσματα που να αφορούν όχι μόνο μία ουσία, αλλά όλες τις ουσίες μιας συγκεκριμένης ομάδας. Όπως είπα, αυτή την ε, απλούστευση θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε από τον χρόνο και είμαστε ο πρώτος οργανισμός παγκοσμίω που έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο και όπως είπα, γι' αυτό το σκοπό αναδιοργανώμαστε πλήρως για να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας. Πάμε στις ε, ε, αδειοδοτήσεις έχουμε διάφορες, ε, διάφορα υποκατάστατα. Να σας πω ότι γενικά ότι η αδειοδότηση είναι ένα νέο σύστημα, σχετικά νέο, αν το συγκρίνουμε τα αδειοδοτήσεις των περασμένων ετών. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά. Να σας πω όμως ότι και όλοι οι φορείς, όλοι οι συμμετέχοντες ε, στην Ευρώπη γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα σύστημα διοδότηση το οποίο μπορούν να συμβάλλουν. Τι κάνουμε εμεί ε, σε θέματα ε, εναλλακτικών λύσεων. Έχουμε ε, διευκρινίσει πολύ καθαρά ποια είναι η δική μα δουλειά και ποια είναι η δουλειά τη Κομισιόν, τόσο όσον αφορά τα υποκατάστατα ή τι εναλλακτικέ, όσο και σε θέματα κοινωνικο-οικονομική ανάλυση. Και όσον αφορά τα συμπεράσματα του κατά πόσο μπορεί να χορηγηθεί ε, αδειοδότηση ή όχι, όλα αυτά βρίσκονται στο Στι αρμοδιότητες της Κομισιόν. Και όλα αυτά τα αναφέρουμε στι γνωμοδοτήσεις μας, ε, ώστε να μπορέσει η Κομισιόν να λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Προφανώς, οι γνωμοδοτήσεις ή οι αποφάσεις της Επιτροπής σήμερα βασίζονται σε παλιότερε δικέ μα γνωμοδοτήσει. Συνεπώ, ε, δεν έχουν ακόμα αυτή τη νέα μορφή. Αλλά όταν ε, θα τελειώσει αυτό το κύμα των γνωμοδοτήσεων και θα έχει περάσει μέσα από την Κομισιόν, εγώ προσδοκώ ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο εξάμεινο του χρόνου που θα έχει συμβεί αυτό θα δούμε και τις, θα φανεί και που εκδίδονται από την Κομισιόν. Αλλά έχουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ ημών και της Κομισιόν όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, στην ιστοσελίδα μας και συζητώντα με επιχειρήσεις προωθούμε ιδιαίτερα τα υποκατάστατα, τις εναλλακτικέ ε, συζητάμε με όλους τους ετούντες όσον αφορά την ανάλυση των αναλλακτικών ουσιών και θεωρούμε ότι φέτος η κατάσταση βελτιώνεται ως, όπως είπα, στην περίπτωση του χρωμίου αυτή η αντικατάσταση με το χρώμιο 3 και κάποιες άλλες καινοτόμες τεχνολογίες είναι κάτι που προέκυψε κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Και φυσικά θέλουμε αυτό να γίνεται πριν εμείς εκδώσουμε γνωμοδοτήσεις στην ΕΚΑ. Οπότε πρέπει να διαδώσουμε την καλή αυτή είδηση σε όλη την Ευρώπη και αυτή η παραγωγή εναλλακτικών ουσιών, εναλλακτικών χημικών να ε, δηλώνονται σε εμά πιο νωρί. Οπότε έχουμε ακόμα πολλή δουλειά, πολύ περιθώριο βελτίωση, αλλά κάποιε βελτιώσει είναι ήδη ερωτέ. Για το χρώμιο 6 ειδικότερα θεωρώ ότι αξίζει να σημειωθεί πω όλε οι γνωμοδοτήσει που έχουμε εκδώσει εμεί Ε, εκεί βλέπουμε ότι όλες οι εταιρείε που ζήτησαν εξουδότηση ε, του ζητήθηκε να διατηρούν ε, τιμή 2 ppm ε, στο χώρο εργασίας. αυτή είναι κάτω από την ανώτατη τιμή έκθεσης. οπότε η εξουδότηση παρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζομένους από ότι έχουμε ως όριο έκθεση στον εργασιακό χώρο. Οπότε είναι συμπληρωματικά όλα αυτά και συνεργάζονται πολύ καλά μαζί για την προστασία των εργαζομένων. Πάμε στους περιορισμούς. Εδώ έχουμε το ζήτημα των ελαστικών και βραχυπρόθεσμα φυσικά πάντα γίνεται συζήτηση για τα παραδοσιακά χημικά που απαγορεύονταν ως πρωτεύοντα υλικά αλλά επανέρχονται ως δευτερεύοντα υλικά στην οικονομία. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εμείς να αξιολογήσουμε στον οργανισμό μας αλλά και που πρέπει να αποφασίσουν ε, οι υπευθυνοί χαρακτήρες πολιτικής κατά πώ θέλουν να έχουν χαμηλό επίπεδο προστασίας αν θα αποδέχονταν υψηλότερα η περιεκτικότητα ε, παλιών χημικών ε, ως δεύτερου υλικού από ό,τι αποδέχονταν ως πρωτεύων υλικό. Φυσικά αυτό δημιουργεί στρέβλωση στην οικονομία, αλλά από την άλλη προωθεί και την, και την ανακύκλωση. μικροπλαστικά. Εκεί θα το πω πολύ καθαρά όσον αφορά την ορολογία. Η γραμματεία της ΕΚΑ έχει εκδώσει μια πρόταση περιορισμού που σταδιακά καταργεί τη χρήση των μικροπλαστικών σε όλες τις χρήσεις όπου βρίσκονται στην Ευρώπη. Αυτή η πρόταση συζητείται στην Επιτροπή Εξολόγησης Κινδύνου της ΕΚΑ και αναμένουμε η γνωμοδότηση να ολοκληρωθεί στην Επιτροπή Εξολόγησης Κινδύνου και στην Επιτροπή Κοινωνικού Οικονομικής Ανάλυσης του χρόνου, ούτως ώστε μετά να μπορέσουν να περάσουν να περάσει γνωμοδότηση στην Επιτροπή για να εκδώσει την εκτελεστική απόφαση κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτό ή όχι, ανάλογα με τη δική μα γνωμοδότηση βάσει τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων. Θα έχουμε ολοκλήρωση, λοιπόν εντό τη 15 μήνης προθεσμίας Ποιο χρονοδιαγράμμα μπορούμε να αναμένουμε. Να ζητήσω από τους συναδέλφους μου αν δεν πω κάτι να το ελέγξετε και να το ξαναπούμε πότε αναμένουμε τη γνωμοδότηση Α, μου το στέλνουν. June. Τον Ιούνιο του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. So, June we our and hand... τον, Ιούνιο, Ιούνιο λοιπόν θα ολοκληρώσουμε την εργασία μας και θα καταθέσουμε τις γνωμοδοτήσεις μας στην Επιτροπή ώστε να λάβει αποφάσεις μέρος της ανάλυσης εστιάζει και σε εναλλακτικέ για τα μικροπλαστικά και συνεπώς εξετάζει τον χρόνο που χρειάζεται για την εφαρμογή των εναλλακτικών και αυτό είναι ένα εργαλείο έτσι ώστε να προωθήσουμε την χρήση εναλλακτικών και τον εντοπισμό εναλλακτικών που είναι πιο ασφαλής. Τώρα, πάμε στα σχόλια ε, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, συμφωνώ. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά σημεία και των δύο τομέων, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες, συνεργασίες για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους με χαμηλότερο κόστος για τον εργοδότη. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες. Τα όρια έκθεση στην εργασία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, σημαντικό εργαλείο. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα, και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ώστε να βελτιωθούμε. Στόχος είναι να υπάρξει συζήτηση και δέσμευση και από τις δύο πλευρές. Και όταν ε, μιλώ για δέσμευση δεν αναφέρομαι τόσο σε κάτι το πολιτικό, όσο σε ένα επίπεδο πιο τεχνικό δέσμευσης. Τα καλλιτικά τώρα. Δεν συμφωνώ στο ότι ο κανονισμός REACH υπονομεύει τον κανονισμό για τα καλλιντικά και την απαγόρευση της χρήσης σε ζώα και της δοκιμής σε ζώα. Θεωρώ ότι πρόκειται για δύο συμπληρωματικά νομοθετήματα και ότι γίνεται σεβαστή η απαγόρευση της δοκιμής σε ζώα στον κανονισμό REACH και σε άλλους σχετικούς κανονισμούς Στόχος είναι να διασφαλίσουμε την υγεία των καταναλωτών ε, σε άλλα κομμάτια και όχι μόνο στα καλλιντικά. Είναι πιο γενική αυτή οι κανονισμοί. Υπάρχει λοιπόν κάποιες φορές μία διάσταση ανάμεσα στην πολιτική βούληση να μην υπάρχει ε, καθόλου, να μην υπάρχει καμία δοκιμή σε ζώα για τα καλλιντικά σε σχέση με τις διατάξεις του, REACH, ε, του κανονισμού REACH και την χρήση χημικών από τους εργαζομένους. Πράγματι έχετε δίκιο ότι η γραμμή αυτή είναι πολύ λεπτή, αλλά είναι πολύ καλά καθορισμένη. Είναι πολύ καλά καθορισμένο πότε χρειάζεται δοκιμή υπό τον κανονισμό REACH και πότε υπό τον κανονισμό για τα καλλιντικά. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Εμπορίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν έχει υπόσταση εκτός Ευρώπης όταν βρισκόμαστε στη ΣΚΟΠ ή οπουδήποτε αλλού, βρισκόμαστε πίσω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπούμε τεχνικά την Επιτροπή. Άρα λοιπόν δεν συμμετέχουμε σε κάποια εμπορική συμφωνία άμεσα. Μέσω των συνεργαζόμενων υπηρεσιών μας λαμβάνουμε ερωτήσεις, αλλά εκεί τελειώνει το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, αναθεώρηση του REACH και γενικά την χημική βιομηχανία. Πολύ συχνά αναφέρεται ότι θα πρέπει στα σύνορα να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε τις παράνομες εισαγωγές διαδραματίζουμε και εμεί ένα ρόλο σε ό,τι αφορά το συντονισμό και τη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και όπως είπα προηγουμένω, αυτό είναι κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε ώστε να αυξήσουμε τις προσπάθειες και την εργασία σε αυτό το τομέα. Φυσικά η δική μας η δουλειά είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι τη συνολική ανάγκη που υπάρχει να εφαρμοστεί η νομοθεσία στα σύνορα σε ό,τι αφορά το διοξίδιο του Τανίου. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα που θέσατε. Δεν είμαι προετοιμασμένος. Δεν έχω διαβάσει με λεπτομέρειες την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου. Πρόκειται για τεχνικές σημειώσεις ε, με βάση ένα συγκεκριμένο παράρτημα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, αλλά φυσικά θα μπορούσα να σας δώσω μια γραπτή απάντηση συνεργασία με τους συναδέλφους μου. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο διαδραματίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο που αναφέρεται στις συνθήκες. Ο δικός μου ρόλος είναι να εξετάζω κατά πόσον υπάρχουν ψηφίσματα που έρχονται σε αντίθεση με επιστημονικές γνώμες, γνωμοδοτήσεις που εκφράζουμε από την πλευρά της ΕΚΑ. Και διαβάζοντας εδώ αυτά τα έγγραφα βλέπω ένα κομμάτι της ιστορίας και όχι την πλήρη εικόνα. Αυτό που βλέπω λοιπόν εγώ από τη δική μου την πλευρά είναι ότι η ΕΚΑ πιστεύει ότι το διοξείδιο του τιτανίου είναι καρκινογόνο διαεισπνοής εμπίπτει στην κατηγορία 2, δεν εμπίπτει στην κατηγορία 1α1β, αλλά θεωρούμε ότι ανήκει στην κατηγορία των καρκινογόνων διαεισπνοής 2. Τα επιστημονικά στοιχεία το αποδεικνύουν αυτό και μπορώ να σας πω πού προέρχονται τα στοιχεία μας. Προέρχονται από το παγκόσμιο σύστημα ε, GHS και από την Επιστημονική Επιτροπή που εξετάζει αυτό το ζήτημα. Τα στοιχεία που εξετάσαμε είναι τα στοιχεία που η βιομηχανία θεωρεί ότι πληρούν τα κριτήρια του ΡΙΤΣ και με βάση αυτά τα στοιχεία η Επιτροπή ΡΑΚ θεωρεί ότι το στοιχείο αυτό είναι ε, καρκινογόνο ε, διαεισπνοής ε, κατηγορίας 2. Τώρα, αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην αρέσουν στη βιομηχανία, αλλά πριν από κάποια χρόνια η βιομηχανία μας είχε καταθέσει αυτά τα στοιχεία σε σχέση με το θέμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα στοιχεία, όπως σας είπα και προηγουμένως, θεωρούμε ότι είναι καρκινογόνο διαεισπνοής. Η ΕΚΑ έχει αρμοδιότητα διαχείρισης κινδύνου και προφανώς το να θέσουμε όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας είναι μια επιλογή και πολύ σύντομα θα σας εξηγήσω το ζήτημα της ταξινόμησης. Ο λόγο που κάνουμε την ταξινόμηση είναι όταν ένα εργαζόμενο πιάνει κάποιο χημικό να βλέπει την ετικέτα και να γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο χημικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η ετικέτα ώστε ο κόσμο να προσέχει, οι εργαζόμενοι να το προσέχουν και να το χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν όλα μα τα εργαλεία, τα νομοθετικά εργαλεία βασίζονται στην επικοινωνία έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι είναι αυτό που χειρίζονται δεν έχει να κάνει τόσο με την ταξινόμηση όσο με το να θέτουμε ε, όρια έκθεσης. Το, η τοποθέτηση ορίων έκθεσης είναι ως εξής. Είναι σαν να έχουμε έναν δρόμο με πάρα πολλές στροφές, να έχει 30 χιλιόμετρα όριο κυκλοφορίας ε, ταχύτητας, ώστε να μην υπάρχουν ε, ατυχήματα, χωρίς να έχουμε καμία πινακίδα. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και με αυτά τα όρια. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο, να υπάρχουν και ετικέτε αλλά και τα όρια έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να αναγνωρίσουν αυτέ τι ουσίε. Αυτέ είναι κάποιε αρχικέ μου σκέψει και ξέρω ότι μετά φυσικά το ζήτημα αυτό θα το συζητήσετε και αργότερα. Σας ευχαριστούμε αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να μας το πείτε πριν από αύριο που είναι ψηφοφορίες. Ε, λοιπόν, ε, τώρα, από του εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβούλιο, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια σχόλια. τους Ρουμπενευρά και το η κυρία Κριστέλ Μπερνάρτ. Ε, ναι, ευχαριστώ. Σημείωσα τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Ε, δεν πρόκειται τώρα να μπω στη διαδικασία του να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα. Ε, ήταν το πρώτο μου έτος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Μάλλον θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία τα οποία με απασχολούν. Πρώτα απ' όλα σημείωσα ότι η ΕΚΑ προσπαθεί να δράσει γρήγορα με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα τα στοιχεία που έχει στη θέσή τη στα του στρατηγικού σχεδίου. Ε, προσπαθεί να, κατανέμει τους πόρους, τη παρογνωμοσύνη που υπάρχει, να ακολουθεί τις κατάλληλες διαδικασίες ε, για να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική στην διεκπαιρέωση των καθηκόντων. Διάδοθηκαν κάποια παραδείγματα. Ε, όλα αυτά βεβαίω εγκρίνονται στη συνέχεια από το, από το Συμβούλιο το Διαχειριστικό. Ε, δύο σημεία τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν προκλήσεις επανέρχομαι στις συνεδριάσεις του, του Συμβουλίου. Το πρώτο έχει να κάνει τον προπολογισμό. Ε, η ΕΚΑ, όπως ξέρετε, έχει έναν προπολογισμό κειμενόμενο. Ε, έχουμε βέβαια κάποιες προβλέψεις ό,τι αφορά τα έσοδα από τα τέλη, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι. Γι' αυτό τα διάφορα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει είναι πάντα λίγο μετέωρα. Ε, αν ιδιαίτερα να προσθεθούν και άλλα καθήκοντα, χωρίς να μας δοθούν πόροι, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Και μια άλλη πρόκληση είναι ότι η ΕΚΑ είναι μια ψηφιοποιημένη σε μεγάλο βαθμό ε, υπηρεσία, διαθέτει πολλούς πόρους ε, για την βάση δεδομένων, την ανταλλαγή πληροφοριών, είναι συγκεκριμένες ε, και οι προθεσμίες και ελπίζουμε ε, να συνεχίσουμε να τηρούμε τις προθεσμίες αυτές ε, ε, παρά τις προκλήσεις που έχουμε να δημιουργήσουμε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται αυτός ο ετήσιος διάλογος όπως είπατε και εσείς. Βεβαίω θα υπάρξει μια νέα στρατηγική για μηδενική μόλυνση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Green Deal. Οπότε η πραγματογνωμοσύνη σας θα είναι σίγουρα καλοδεχούμενοι τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και έτη. Θα τα πούμε λοιπόν σύντομα ξανά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε και σας και την ομάδα σας για όλα όσα, έχετε, όλα όσα έχετε κάνει. So we move to the other agenda item. Uh, Πάμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξη, στο σημείο 6, ε, με την αντίρρηση. Με βάση τον κανόνα 113, ε, για την συσκευασία, ε, την ε, ετικετοθεσία σχετικά με το δεξίδιο του Τιτανίου. Παρακαλώ το λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια. Ναι, συγγνώμη, πόσο χρόνο έχω, ρωτάει η κυρία Ζαλεύσκα. Τέσσερα λεπτά. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αυτή η συζήτηση για το διοξίδιο του τιτανίου έχει ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να πω ότι ο κ. Χάνσελ προηγουμένω δεν με έπεισε. Βέβαια, δεν είναι θέμα πεπιθήσεων. Είναι θέμα πολιτικών στοιχείων. Εγώ, αφού ανέλησα όλα τα στοιχεία, έχω μία αντίρρηση ε, είμαι κατά για το καλό του περιβάλλοντος, για το καλό των καταναλωτών, των συμπολιτών μας. Διαπιστώνω ότι η συζήτηση κρατάει εδώ και δύο χρόνια. Ε, δεν έχουν προκύψει κάποια νέα στοιχεία. Η Κομισιόν δεν έχει διαθεσή της τέτοια στοιχεία. Έχει γίνει μια μελέτη εξαιρετικά κοστοβόρα και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα εκείνης της μελέτης μπορούμε να τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους. Ενώ η δοκιμή έγινε πάνω σε ε, ε, ποντίκια. Εδώ μιλάμε βέβαια για κατηγοριοποίηση, για ταξινόμηση. Θέλουμε να αλλάξουμε κατηγορία α, για αυτό το προϊόν, δηλαδή να πούμε ότι είναι καρκινογόνο. Στα πλαίσια της συζήτησης βέβαια για την υγιεινή στο χώρο εργασίας και για την ασφάλεια στο χώρο εργασία. Γιατί, διότι τις περισσότερες φορές αυτή η ουσία έχει τη μορφή ε, πούδρας, σκόνης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτήν την ε, ουσία στα πλαίσια της οδηγίας που έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας και από εκεί και πέρα έχουμε μία κατάσταση όπου κάποιοι άνθρωποι δεν ε, εκτίθενται ε, στο διοξείδιο του Τανίου με τον ίδιο τρόπο που εκτίθεται σήμερα. Επίσης δεν μπορούμε να δεχτούμε ελήψη μελετών αυτή την ιδέα να αλλάξει ε, κατηγορία. Διότι το διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται για χιλιάδες προϊόντα και δεν υπάρχει κάποια μελέτη ή κάποιο στοιχείο που να μας ε, επιβεβαιώνει ε, τους ε, κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων. Επίσης, το διοξείδιο του τιτανίου έχει κάποιες ιδιότητες ιδιαίτερες, ιδιαίτερα όταν είναι σε επαφή έχει σε επαφή με το δεξίδιο του θείου, δεν έχουμε νέα στοιχεία, δεν έχουμε καινούριε αναλύσεις, δεν υπάρχουν καθόλου επίσης οικονομικές μελέτες που να ε, μας λένε ποιο θα είναι το κόστος αντικατάστασης αυτής της ουσίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, πραγματικά, εγώ είμαι κατά αυτού του σχεδίου. Θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τις συνθήκες εργασίας, να δούμε την οδηγία για τις συνθήκες εργασίας, εργασιών, που ενδεχομένως πρέπει να τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Να δο... διαρθρώσουμε κάπως τη συζήτηση με βάση τις πολιτικές ομάδες, ξεκινώντας με το ΕΛΚ. Ποιος θα πάρει το λόγο για το ΕΛΚ. Ο κ. Σπυράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ε, εξηγήσω επί της αρχής. Δεν είμαστε κατά της ταξινόμησης του διοξιδίου ε, του τιτανίου, αλλά ως ΕΛΚ θεωρούμε ότι η ταξινόμηση ως πιθανό καρκινογόνο δημιουργεί αβεβαιότητα και ίσως έχει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορες βιομηχανίες και επίσης στην υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η ταξινόμηση αυτή θα επιβληθεί μόνο σε σκόνη που περιέχει 1% ή παραπάνω διοξείδιο του τιτανίου. Ωστόσο η πούδρα ή η σκόνη δεν ορίζεται και άρα υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και αυτό μπορεί να επηρεάσει project, έργα τα οποία μπορεί να, μπορεί να ε, συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία και κατανοώ ότι έχουν γίνει δοκιμές σε πειραματόζωα, σε ποντίκια και από την άλλη χρειάζεται πολύς χρόνο έτσι ώστε οι μελέτες να φτάσουν σε ασφαλή ε, συμπεράσματα. Ψηφίζουμε υπέρ λοιπόν της αντίρρησης Φυσικά αναμένουμε από την Επιτροπή να μας δώσει επιπλέον πληροφόρηση ε, για την ε, πρόταση που έχει καταθέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Δεν είναι εδώ λοιπόν η εκπρόσωπος. Αυτό που μπορώ όμως να πω είναι ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες δεν υποστηρίζουν την αντίρρηση. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί, αλλά αυτή είναι η δική μας η θέση. Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι. Σίγουρα βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Ωραία. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ ε, βεβαίως δεν είναι ενωμένη η ομάδα μα η Renew. Ε, η ομάδα μας πάντως είναι κατά της ε, αντίρρησης. Ε, με επιχειρήματα σύμφωνα με την οποία υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να υπάρξει προστασία. Ε, εγώ προσωπικά επειδή προέρχομαι από το κόσμο της βιομηχανίας ε, δεν συμφωνώ με αυτά που ο πρόεδρος της ΕΚΑ. Υπάρχει κατάρτιση για τους εργαζομένους. Ε, αν δεν έχουν καλή κατάρτιση θα υπάρχει πρόβλημα. Ε, διαπιστώνω ότι εδώ δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε το κατά πόσο είναι τοξικό το προϊόν ή όχι, αλλά το κατά πόσο υπάρχει ένας τρόπος για να υπάρξει βιωσιμότητα. Και αυτό μέσω αυτού το, μπορεί να γίνει μέσω του ορίου σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας. Ε, αυτό μπορεί να βοηθήσει ε, σε ό,τι αφορά αυτούς που εργάζονται στον τομέα αυτών και βεβαίως μιλάμε για σκόνη σε με μεγάλη ε, περιεκτικότητα ε, και με μεγάλη και μακροσκελή έκθεση. Ε, δεν μιλάμε για το προϊόντα το οποίο μοιράζονται στους πολίτες. Οπότε εμείς δεν είμαστε κα, υπέρ μάλλον αυτής της αντίρρησης. Δεν συμφωνούμε με την αντίρρηση. Ευχαριστώ για τους πράσινους τώρα. Η κυρία Πάρης, ε, ναι, ευχαριστώ. Μου κάνει εντύπωση διότι ε, βλέπω ότι το ΕΛΚΑ πραγματικά θέλει να δώσει, λέει ότι θέλει να δώσει μάχη κατά του καρκίνου και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή έχετε αντίρρηση για μια επισήμανση για προϊόντα τα οποία είναι καρκινογόνα. Εδώ υπάρχει αντίφαση. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία, όπως είπαν κάποιοι. Όπως είπε ο κύριος Χάνσεν, Έχουμε την αξιολόγηση της ΕΚΑ, έχουμε την αξιολόγηση της IIA, IIRC, μάλλον πάει προς την ίδια κατεύθυνση, είναι μια καρκινογόνος ουσία και θέλουμε μια επισήμανση που να αναφέρει απλώς ε, να το αναφέρει αυτό, έτσι ώστε και οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτέ να έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε για να μπορέσουμε να του προστατεύσουμε. Να μην ψεκάζεται, να λέει απλώ μια επισήμανση, τίποτα άλλο. Ε, δεν θέλει κάποιο λόγο για την ομάδα ID. Ε, ECR. Α, για την ID. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η θέση μας είναι αυτή την οποία έχουμε αναφέρει εδώ και καιρό και την γνωρίζετε για τα καρκινογόνα. Δεν είμαι βέβαιη ότι με μία αντίρρηση ε, έχει νόημα να αρχίσουμε να συζητάμε και να ε, Αφιζητούμε τους κανόνες που ισχύουν για την ε, επισήμανση και την επαναξιολόγηση των προϊόντων. Όλα αυτά πρέπει να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, όσο γίνεται με την προστασία των εργαζομένων. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές ε, τους στόχους τους, ε, αλλά αυτό που ισχύει, αυτό που, πρωτεύει είναι η προστασία των εργαζομένων και αυτή δεν εξασφαλίζεται με αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστώ κυρία Χάζενκαμπ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα για την κατηγοριοποίηση του διοξιδίου του τιτανίου ως καρκινογόνο. Υπάρχουν ε, και ουσίες που έχουν μείνει εκτός από αυτή την κατηγοριοποίηση που, έχουν διοξείδιο του τιτανίου και που είναι υγρής μορφής. Και υπάρχει πρόβλημα με τον κανονισμό αυτό. Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμβιβαζόμαστε απέναντι ε, σε κάποια οικονομικά αιτήματα. Πρέπει εδώ να ισχύει το πιο υψηλό επίπεδο κατηγοριοποίησης ε, και ταξινόμησης ε, για αυτά τα καρκινογόνα. Χρειάζεται μια πιο ισχυρή στρατηγική αντικατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τη χάνει δημοκρατική υποστήριξη ούτε από τα κρατημέλη, ούτε από το Κοινοβούλιο, για να επιτρέψει, παραδείγματο χάρη, τα Βεβαίω, ε, εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνώμη της Επιτροπής ε, Αξιολόγησης Κινδύνου. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτή την αντίρρηση, την οποία, όπως ξέρετε, την έχει γράψει ένα λόμπι Πέτρε Λίζ είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς ως ΕΛΚΑ, σαφώς κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με αυτό, θέλουμε να καταπολεμάμε τον καρκίνο. Αυτό θέλουν και οι πράσινοι. Το ίδιο θέλουμε και εμείς. Αλλά ε, θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με απόλυτη ακρίβεια και εγώ συζήτησα πρόσφατα με το Γερμανικό Κέντρο για τον Καρκίνο και υπάρχουν πάρα πολλά καλά απορίσματα για τις αιτίε ε, του καρκίνου και τα χημικά που συζητάμε ε, το, κέντρο, το Γερμανικό Κέντρο του Καρκίνου δεν μπορεί να μας παρουσιάσει συμπεράσματα. Υπήρξε μία περίπτωση. Η συνάδελφος κυρία Σπυράκη έκανε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε τα συγκεκριμένα σημεία, αλλά το θέμα είναι ότι στη Γερμανία ο οργανισμός που ασχολείται με την προστασία των εργαζομένων λέει ότι ο κανονισμός είναι περιττός. Έχουμε επαρκείς κανονισμούς για να προστατεύουμε επαρκώς τους εργαζομένους και ο υπουργό Εργασίας των Σοσιαλδημοκρατικών λέει το ίδιο. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο. Αυτή τη στιγμή μα βοηθά πραγματικά αυτό. Εγώ έχω τρει συγκεκριμένε ερωτήσει προ την Κομισιόν. Πρώτον, είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι υπάρχουν ε, ε, παραδείγματα μόνο σε τροκτικά. Υπάρχουν ε, πορίσματα για ανθρώπους και αν υπάρχουν μπορείτε να μας τα στείλετε. Δεύτερον, στο σημείωμα που έστειλε η Κομισιόν λέγει ότι η τα αποτελέσματα για την ανακύκλωση είναι ελάχιστα, αλλά ποια είναι αυτά σε περίπτωση που προκύψουν. Και τρίτον, τι ακριβώς ε, επισημαίνεται με επισήμανση. Αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο χρώμα, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά τι γίνεται ε, ο, άμα ε, υπάρχει, υπάρχει κάτι το οποίο στην όλη διαδικασία προκαλεί καρκίνο. Θα πρέπει να γνωρίζουν τι κάνουν οι εργαζομένοι. Και κάποια υποκατάστατα επίση θα μπορούσαν να δημιουργούν προβλήματα. Ποιε ακριβώ λύσει προτείνονται. Thank you, sir. I will give the floor. Uh, Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος για να κλείσουμε αυτή την ε, συζήτηση για το διοξίδιο του Τιτανίου. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε που μας κάλεσατε εδώ να συζητήσουμε αυτή την αποφασή μας να το ε, κατηγοριοποιήσουμε ως καρκινογόνο κατηγορίας 2, το διοξίδιο του Τιτανίου. Όπως ξέρετε, σκοπός του κανονισμού είναι να παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας ε, για την υγεία και το περιβάλλον, προσδιορίζοντας τους κινδύνους βάσει των ιδιωτήτων των ουσιών. Υπάρχουν δύο τρόποι κατηγοριοποίησης ή ε, είτε αφήνουμε τη βιομηχανία να κάνει ταξινόμηση ή κάνουμε εναρμονισμένη ε, κατηγοριοποίηση είτε με πρωτοβουλία των κρατών μελών είτε με πρωτοβουλία της βιομηχανίας. Ο σχετικός κανονισμός ε, λέει ότι για διαδικασίες καρκινογόνες και για την κατηγορία 2 απαιτείται εναρμονισμένη ταξινόμηση. Η πρόταση λοιπόν, η απόφαση που λάβαμε βασίστηκε στην ε, Επιτροπή Αξιολόγηση στην ΕΚΑ. Ξέρετε, Επιτροπή που εξετάζει τι προτάσει των κρατομελών τη βιομηχανία. Και επειδή η Επιτροπή Αξιολόγηση Κινδύνου εξέδωσε την γνωμοδότησή σα, όπω είπαν κάποιοι από εσά πολύ σωστά, από τότε που, που εκδόθηκε αυτή η γνωμοδότηση, κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αφισβήτησε την απόφαση τη Επιτροπή. Το μόνο που έχουμε λοιπόν τεκμήριο είναι αυτή η γνωμοδότηση. Όπως είπα, λοιπόν, η γνωμοδότηση ε, αυτή υπήρξε και ευθυγραμμίστηκε με τα συμπεράσματα του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο, που είναι οργανισμός ε, του ΠΟΕ του ΠΟΗ, συγγνώμη, που είπε ότι το διαπίστωσε ότι το διοξείδιο του τανίου είναι πιθανό καρκινογόνο για του ανθρώπου. Και επίση ευθυγραμμίστε με όλα τα μέτρα τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσαν την απαγόρευση τη χρήση του διοξιδίου του τανίου σε οποιαδήποτε μορφή σε ε, καλλιτικά. Οπότε θεωρούμε ότι η αποφασή μας βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Να σχολιάσω το ζήτημα του κατά πόσο η επισήμωση η στην συσκευασία είναι καλύτερη επιλογή σε σχέση με την νομοθεσία προστασίας. Αυτά τα δύο νομοθετήματα είναι συμβατά είναι ε, και συμπληρωματικά μεταξύ τους. Η εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιαστικά υποχρεώνει τη βιομηχανία να παρέχει ε, πληροφορίες ασφαλείας ε, που προσδιορίζουν την ουσία και που δίνουν οδηγίες στους εργαζομένους για να χειρίζονται ασφαλώς την ουσία. Οπότε αυτή η υποχρέωση του να υπάρχει αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο ε, έχει τα αποτελέσματα προστασία που απαιτούνται. Επίση, ε, η εναρμονισμένη προστασία ε, βοηθά στον ορισμό των ορίων βάσει του σχετική νομοθεσία προστασία. Πρέπει να ξέρουμε όμω ότι το διοξίδιο τιτανίου δεν είναι μόνο επικίνδυνο όσον αφορά του εργαζόμενου. Είναι επικίνδυνο και για τους αυταπασχολούμενους που δεν καλύπτονται από την προστασία την σχετική νομοθεσία προστασίας και μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τους καταναλωτές που εκτίθενται στην ουσία αυτή όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχει εναρμονισμένη ταξινόμηση, θα βελτιώσει την ενημέρωση για την επικίνδυνοτητα της ουσίας και θα βοηθήσει στην ενημέρωση ε, όταν κάποιος ε, πρόκειται να χειριστεί την ουσία. Επίσης επιτρέπει την υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας για την ουσία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εναρμονισμένη ταξινόμηση βασίζεται μόνο στις ιδιότητες ε, και στην επικινδυνότητα της ουσίας και δεν ε, λαμβάνει υπόψη την ε, επικινδυνότητα λόγω έκθεσης. Κάποιοι από εσάς αναφερθήκατε στο γεγονός ότι η σκόνη είναι ασαφής έννοια και θα έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι συστήθηκε η ουσία να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος ε, ε, κατηγορίας 2 με όσφρηση. Ε, στην Κομισιόν ταξινομείται σε μορφή σκόνης με διάμετρο ίση μικρότερη από 10 μικρό χιλιοστά. Οπότε έχουμε συγκεκριμένη διάμετρο σωματιδίων που θεωρείται ότι αυτά αντιστοιχούν στα σωματίδια που μπορεί κανείς να λάβει να, μέσω όσφρηση, Οπότε αυτό βοηθά στην εφαρμογή της απόφασης. There was a question whether the, um, we only had uh, studies on animals. Indeed, we had uh, Διασπνοή, συγγνώμη. Έχουμε και μελέτες ε, ε, στα ζώα που ανέφερα προηγουμένως που παρέχονται από τη βιομηχανία και η σχέση αυτή μεταξύ των αποτελεσμάτων των μελετών σε ζώα και ε, δυνατοτήτων αναγωγής σε ανθρώπους. Γι' αυτό αποφάσισε να μην αποφασίστηκε να μην ταξινομηθεί ως ε, καρκινογόνο, να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο 2. Ε, Η σχέση αυτή μεταξύ των μελετών ε, σε ζώα, των πειραμάτων σε ζώα και των υποθέσεων για τους ανθρώπους οδήγησε σε αυτή την απόφαση της Επιτροπής. Ρωτήθηκε επίσης τι επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση στις ουσίες όπως και στα μείγματα που ταξινομούνται. Μιλάμε για τα μείγματα σε μορφή σκόνης. Κάποια μείγματα δεν θα χρειάζεται να ταξινομούνται σύμφωνα με τη δική μας απόφαση. Θα είναι τα υγρά μείγματα, αλλά θα πρέπει να φέρουν επισήμανση. Δεν θα ταξινομούνται ωστόσο, αλλά θα πρέπει να επισημένονται και να εξηγείται ότι περιλαμβάνουν σωματίδια που μπορούν να προσληφθούν μέσω εισπνοής. Οπότε θα υπάρχει μια υποδοποίηση που θα λέει επικίνδυνο ε, κατά τη χρήση παρακαλούμε μην εισπνέετε. Για εκεί, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση. I think that's replying all the questions that you had. Just to... Απάντηση για τις άλλες ερωτήσεις. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου για τις ερωτήσεις που είχατε. Τώρα να πούμε για την νέα κομισιόν που αναλαμβάνει καθήκοντα σήμερα. Η μάχη κατά του καρκίνου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να προσδιορίσουμε τις ουσίες που προκαλούν τον καρκίνο και χωρίς την ταξινόμηση δεν θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ουσίες ασφαλώς. Thank you very much. So, <clears throat> we will vote, uh, Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε τώρα για αυτό το πολύ... Θα ψηφίσουμε αύριο μάλλον για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Πάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Αντίρρηση σχετικά με τις εισαγωγές τροφών για ζώα συντροφιάς από την Σαουδική Αραβία. Θα δώσω το λόγο στην Ζωέλ Μελίν από το ID. Oui, merci, monsieur. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσω μιας ε, έτσι πολύ μινιμαλιστική ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πράξη του έτσι προτείνει να προσθεθεί και η Σαουδική Αραβία μεταξύ των τρίτων χωρών όπου ε, τα μεταποιημένα τρόφιμα από πουλερικά μπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξηγώντα ότι το βασίλειο τη Σαουδική Αραβία ε, έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κατά, τις κατάλληλες εγγυήσεις σε επίπεδο υγειονομικό. Ε, όμως, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για να απορρίψουμε αυτή την πρόταση. Ο πρώτος είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν χρειάζεται αυτές τις εισαγωγές. Ήδη υπάρχει πλεόνασμα, ήδη έχουμε σημαντική δική μας ε, παραγωγή. Ανοίγοντας ε, τις πόρτες της Ευρώπης ε, σε παραγωγές από τρίτες χώρες, αυτό δυσχεραίνει τους δικούς μας παραγωγούς. Ουσιαστικά μειώνονται και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά μας πρότυπα και τα ποιοτικά μας πρότυπα, διότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα μέσα να ε, ελέγχουμε τακτικά ότι οι επιχειρήσεις των τρίτων χωρών σέβονται αυτού του κανόνε και τι προδιαγραφέ. Είναι θέμα λοιπόν τη αρχή τη προφύλαξη. Επίση, επενθυμίζουμε ότι στη Σαουδική Αραβία ισχύει η Σάρια. Δηλαδή, έχουμε σφαγή των ζώων χωρί πρώτερη αναισθητοποίηση. Σκεφτείτε ποιε είναι και οι υγειονομικέ επιπτώσει ουσιαστικά σφάζονται ζώα χωρίς νάρκωση, χωρίς κανένα σεβασμό της ευμερίας των ζώων. Αυτό αναφέρεται στις αρχές ε, τις ευρωπαϊκές. Εμείς είμαστε λαοί που σεβόμαστε τη ζωή των ζώων. Επίσης, τον επικυρώνουμε από τέτοιες αποφάσεις είναι να ανοίγουμε ε, μία σύμπραξη εμπορική με μία χώρα που παραβιάζει Σαφώ τι αρχέ που περασπιζόμαστε Εμεί εδώ. Συχνά του δαχτυλοδείχνουμε για μη σεβασμό του διεθνου δικαίου. Είναι μια χώρα όπου δολοφονούνται ε, δημοσιογράφοι, χρηματοδοτεί τη δημοκρατία, παραβιάζει τα δικαιώματα των γυναικών και τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Για όλου αυτού του λόγου δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ζητούμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να υποστηρίξετε αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Merci Uh, Τώρα, ας ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ από τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ως κοιόδηση συγγήτρια για αυτόν τον φάκελο, Είμαι ενάντια στην αντίρρηση ε, για τις εισαγωγές τροφών για ζώα συντροφής από τη Σαουδική Αραβία για τους ε, κάτωθι λόγους. Οι αρχές του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας μας έχουν διασφαλίσει ότι η χώρα τους πληρεί τις ε, συνθήκες και τα πρότυπα υγείας σε ό,τι αφορά τα πουλερικά και την παραγωγή πουλερικών. Η προσθήκη λοιπόν της Σαουδικής Αραβίας στη λίστα των χωρών από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί και να, διέλθει, να διέλθουν αυτά τα προϊόντα ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο είναι θεμητό. Πληρούνται λοιπόν όλοι οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς κανόνες και η αντίρρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του εμπορίου. Άρα λοιπόν προτείνω να απορρίψουμε την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ξέρω περισσότερα για αυτό το θέμα, οπότε μπορώ ε, να παρουσιάσω τα επιχειρήματά μας η ομάδα μας δεν θα υποστηρίξει την αντίρρηση για τους ίδιους λόγους που προέβαλε το ΕΛΚ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν αρκετές χώρες όπως η Τουρκία, το Μαρόκο, το Ισραήλ, στις οποίες επιτρέπεται να κάνουν εισαγωγές παρότι ακολουθούν την πρακτική της τελετουργικής σφαγής. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των χωρών σε γενικές γραμμές όμως η ομάδα μας θα ήθελε να συζητήσει το κατά πόσον μπορούμε να βελτιώσουμε την ευζοία ε, σε όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες συναλλασσόμαστε. Και εμείς λοιπόν οι Σοσιαλιστέ Δημοκράτες είμαστε ενάντια, ψηφίσουμε κατά της αντίρρησης. Για το Ρηνιού τώρα, η κυρία Στεφανούτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφέρω να αναφερθώ στα ζητήματα αρχής. Είναι ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό. Το θέμα της μεταφοράς των ζώων, και αυτό το έχουμε συζητήσει σε πολλά φόρουμ εδώ ε, στο Κοινοβούλιο. Στη Ρουμανία, από όπου προέρχομαι, ένα μεγάλο φορτίο 14.000 ε, προβάτων πνίγηκε στη Μαύρη Θάλασσα και αυτό είχε να κάνει με μια διεθνή συμφωνία, γιατί από τη στιγμή που κάποιο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, ε, ένα πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, δεν εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και ρωτώ την Επιτροπή, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτέ οι διμερεί συμφωνίε που περιέχουν πρότυπα ευζοία ε, πώ μπορούν να ενσωματωθούν και στι διεθνεί συμφωνίε. Ευχαριστώ. Για του πράσινου τώρα. Δεν υπάρχει κανένας ομιλητή για του πράσινου. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, συζητάμε για ευημερία των ζώων εδώ, για το εύζην των ζώων. Θέλουμε αυτό να το βελτιώσουμε. Ε, όμως συζητάμε και το ψήφισμα, έτσι. Το S&D λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ε, κατά των ε, κρατών, ε, κάποια, κάποια κρατών. Ε, πρέπει να έχουμε να ισχύει για όλες τις χώρες αυτό που υπόθηκε. Παρακαλώ, ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμεί δεν συμφωνούμε με την αντίρρηση όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές. Είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας είπε ότι γίνεται προσπάθεια από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε λόγο να το πιστέψουμε και δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος αυτός να να αντιπαρατεθούμε με την Σαουδική Αραβία, οπότε δεν συμφωνούμε με την αντίρρηση. Θέλει κάποιο το λόγο από την ΚΟΕ. Μάλιστα, δεν θέλετε το λόγο. Πω, ενδιαφέρον. Ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Υγείας, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλό σας απόγευμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού εγγραφιστηγαμίζεται πλήρως ε, με αυτά που προβλέπονται στη βασική πράξη. Μια χώρα μη μέλος της Ένωσης που ζητάει άδεια εισαγωγής προϊόντων ε, ζωικής προέλευσης αξιολογείται πολύ αυστηρά για να εξασφαλίσουμε ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες ε, και παρέχει τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις ε, κατά την των ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα τη ευημερία των ζώων. Είναι πολύ σημαντική η προστασία των ζώων και κατά τη φαγή του. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν το άρθρο 12 του κανονισμού 1019 ε, του 2019 επιβάλλει πολύ συγκεκριμένε προποθέσει για την εισαγωγή κρέατο από τρίτε χώρε. Βεβαίω αυτέ οι απαιτήσει δεν εφαρμόζονται για υποπροϊόντα ε, όπως την τροφή για κατοικίδια ζώα. Ε, υπάρχουν βεβαίως άλλα μέτρα ε, υγειονομικά στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου για αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα, λοιπόν, η τροφή για κατοικίδια ζώα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις προβλέπω το σχετικό κώδικα για την υγεία των ζώων στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ζώων. Βέβαια, ο κώδικας δεν αναφέρει κάποια διάταξη για την ευμερία των ζώων στην περίπτωση των, των, των, των για κατοικίδια ζώα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εισαγωγή από τη Σαουδική Αραβία, εμείς εξολογήσαμε το σύστημα ελέγχου που υπάρχει επί τόπου και θεωρούμε ότι παρέχει τις αγγιήσεις που προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 44 του κανονισμού 1019 του 2019, Υπάρχει μια παρέκκληση λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά ε, την ε, νάρκωση όταν έχουμε μια τελετουργική σφαγή. Πρέπει να σεβαστούμε τις θρησκευτικές παραδόσεις που προβλέπονται όπως άλλωστε αναφέρει το άρθρο 10 των Μελετών Δικαιωμάτων, τη Χάρτη Μελετών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποτυπώνει το σημείο ισορροπία μεταξύ των στοιχείων που έχουν να κάνουν με την ευμερία των ζώων και τη ελευθερία ε, ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Αποτελείται λοιπόν από προϊόντα ε, πουλερικών ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν 57 χώρες που έχουν των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή για ζωοτροφή για κρατική διαζώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, ε, εάν εγκριθεί ε, αυτή η αντίρρηση θα υπάρξει ζήτημα μη σεβασμού των διεθνών προτύπων θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο ενώ εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που βασίζεται σε κανόνες όταν διεθνές εμπόριο. Μάλιστα, θα ψηφίσουμε από αυτές τις αντίρρησεις αύριο. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης και δίνω το λόγο στη Μισελ Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κομφά. Λοιπόν, ε, ε, αυτή είναι μια πρόταση ψηφίσματος ε, για να αμφισβητήσουμε κάποιο μέτρο του εκτελεστικού κανονισμού της Κομισιόν που βασίζεται στην παρακολούθηση τροφίμων που εισάγονται από την Ιαπωνία. Η Κομισιόν άλλαξε λοιπόν το παράρτημα 2 καταργώντας ε, στο εξή τις απαιτήσει σε θέματα αναλύσεων για κάποια προϊόντα και από γεωγραφική άποψη, γιατί τρεις νομοί είναι αυτοί ε, τους οποίους αφορά το ζήτημα, όπου πήγα και εγώ πρόσφατα ε, οι νομοί που μολύνθηκαν μετά από το γεγονότα στη Φουκουσίμα και την κάνει η Κομισιόν, λέει δεν χρειάζεται πλέον δημοματοληψία, δεν χρειάζεται πλέον να λαμβάνουμε μέτρα. Οι Ιαπωνικές αρχές ε, εφαρμόζουν μέτρα, ξέρουν ότι έχουν, ξέρετε ότι έχουν χαμηλότερα επίπεδα από τα δικά μας, ε, προστατεύουν την υγεία τους ε, περισσότερο από ότι Ευρωπαίοι μάλιστα, ήδη στον παρόδο, αλλά χωρίς να μας λέουν ακριβώς γιατί άρουν ορισμένες δειγματοληψίες, ε, γιατί οι νομοί που μολύνθηκαν προβαίνουν σε τέτοιες δράσεις και βάσει ποιων κριτηρίων αποφάσισαν να προτείνουν αυτό τον κανονισμό. Τώρα έχουμε και κάτι άλλο που μας ανησυχεί. Τι ακριβώς αναλύουμε. Ξέρετε, το ατύχημα της Φουκουσίμα είχε... Ε, είχε μεγάλε επιπτώσει για το Κέσιο 134 και 137 και πολλέ μολύνσει τη εποχή σχετίζονταν με το Κέσιο 137, αλλά τίποτα για το τρίτο. Τεράστιε ποσότητε, ξέρετε, είχαν εκκληθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν, ε, να εκλείονται από τα εγκαταστάσεις της Φουκουσίμα γιατί εξακολουθούμε να ε, βρέχουμε τους πυρήνες ε, οπότε τρίτιο, το τρίτιο αυτό περνάει στο νερό, το νερό περιχειρητίνες για το φιλτράρισμα υπάρχουν διάφορες άλλες ουσίες, πλουτόνιο μεταξύ άλλων και υπάρχει μέσα στα δοχεία και έχουμε μέτρα μόνο για το κέσιο 134 και 137 και εμείς ζητάμε να προσθεθούν τα μέτρα για το τρίτιο που έχει χρόνο ζωής 2,5 ε, και για το στροφείο που ε, έχει 10,5 χρόνια επίσης. Επίσης υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα ότι ξέρετε εισάγουμε ρύζι από την Ιαπωνία. Και γιατί εισάγουμε ρύζι από την Ιαπωνία για να το ταΐζουμε τα βρέφη. Ξέρετε, τα όρια για τα βρέφη και το γάλα είναι 50 μπεκερέλα ένα κιλό. Ε, μόνο που εμείς λέμε όπως οι Κινέζοι, οι Κορεάτες, οι Αυστραλοί γιατί να εισάγουμε ρύζι μολυσμένο ακόμα και αν έχουμε 50 μπεκερέλ ενώ μπορούμε να έχουμε 0 μπεκερέλ ε, και σίου για τα παιδιά και τα βρέφη είναι τελείως παράλογο οπότε εμείς λέμε να σταματήσουμε να εισάγουμε ρύζι για τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη. Μετά έχουμε κάτι άλλο που μας ανησυχεί, γιατί ξέρετε την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία ε, ε από την Ιαπωνία και τους ρώτησα απευθείας. Έχουμε εκατομμύρια κυβικά μέτρα αυτή τη στιγμή αποθηκευμένα στα εγκαταστάσει τη Φουκουσίμα σε κοντέινερ και εγώ ζητάω από την Κομισιόν να κάνει κάτι ώστε να υπάρξουν δειγματοληψίε σε αυτά τα εμπορευματοκιβώτια, να μάθουμε τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα κυβώτια, γιατί λένε ότι υπάρχει μόνο τρίτιο. Ωστόσο υπάρχουν και τα άλλα τα προϊόντα ε, σύνδεξης, ε, πλουτόνιο και άλλες ουσίες και κανείς δεν ξέρει Ε, θυμηθείτε ότι σχετιζόταν η Φουκουσίμα και με κάποια μέλη τη κυβέρνηση και δεν κάνουν ότι δεν έχει συμβεί τίποτα και θέλουν να τα ρίξουν όλα στον ειρηνικό. Και όταν του λέω ότι ξέρετε όλα αυτά τα ραδιενεργά στοιχεία δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτά. Εμεί ε, δεν έχουμε μετρήσει για το τρίτιο και πάνε αυτοί να ρίξουν όλα αυτά τα κυβικά μέτρα στον ε, ειρηνικό με αποτέλεσμα τη μόλυνση το, για τα φύκια, για τα ζώα. Ε, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό και εμεί θα πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο. Γιατί ξέρετε, έχουμε τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Ιαπωνία. Γι' αυτό το λόγο σα καλώ να ψηφίσετε υπέρ αυτή τη πρώτη ψηφίσματο ώστε να πιέσουμε την ε, Επιτροπή να αποσύρει τον εκτελεστικό κανονισμό και να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 το αργότερο, ώστε να διασφαλιστεί ε, επαρκέ επίπεδο προστασία τη ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντο. Και επίση για να λάβουμε περισσότερε πληροφορίε για τα όσα συμβαίνουν στην Ιαπωνία και κυρίω για το ποιο λόγο να εισάγουμε μολυσμένα ιαπωνικά προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ για το ΕΛΚΑ. Κύριε Τόπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον εισηγητή του ΕΛΚΑ, ε, τον κύριο Κάνεβο, ο οποίος είναι κατά αυτής της αντίρρησης. Δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Η θέση του βασίζεται στην αξιοπιστία των ελέγχων που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή βάσει των δεδομένων που υποβάλλονται από τις Ιαπωνικές Αρχές για το 2017 και 2018 και τα παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία μη υπέρβασης των ανώτων ορίων ραδιενέργειας σε εξεταζόμενες ζωοτροφές και τρόφιμα για, και για διάστημα μετά από το ατύχημα. Επιπλέον επιχείρημα κατά της αντίρρησης θεωρεί ότι είναι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ιαπωνία. Από αυτή την άποψη θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερες πιο λεπτομερείς πληροφορίες δεδομένων των σχέσεων μεταξύ, στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο οργάνων, αλλά το πρόβλημα αυτό δεν πρέπει να αποδίδεται στις ε, σχέσεις και τις ανταλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας. Και τέλος, ε, ε, κατά συνέπεια το ΕΛΚ θα απορρίψει αύριο αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να πω στην κυρία Ριβαζή ότι αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τα ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι ζωοτροφές και τρόφιμα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρουσιάζουν πρόβλημα. Όσον αφορά αυτέ τι αντιρρήσει, έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, η διαφάνεια των δεδομένων και δεύτερον, νερό ψήξη. Λοιπόν, για τη διαφάνεια των δεδομένων ε, ε, γίνεται η σχετική συζήτηση ε, από τα μέλη. Μετά έχουμε το νερό ψήξη. Υπάρχουν κάποιε απαιτήσει όσον αφορά αυτό το νερό. Τι συμβαίνει με αυτό, τι πρόκειται να συμβεί σε αυτό πριν το 2021. Εγώ θα ήθελα να γίνει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για το νερό ψήξης. Οπότε αυτά εμείς ως σοσιαλιστές δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε την αντίρρηση ακόμη και παρότι ε, συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ε, εμπλακεί σε όλα αυτά ε, στους ελέγχους των υποδομών στη Φουκουσίμα, οπότε δεν θα υποστηρίξουμε την αντίρρηση. Αντιθέτως θα θέλαμε να γίνει κάτι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το Renew η Βερονίκ Τρινό. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Τρίγια Λενόρ, παρότι δεν έχουμε κάποιο περιστατικό μετά από 7 χρόνια ελέγχου και παρότι η συνάδελφος ε, η Μισελ ε, ε, ξέρετε, τα επίπεδα απαγόρευση ε, που αναφέρονται δεν αφορούν όλα τα τρόφιμα και παρότι η απειλή αυτή τη στιγμή όσον αφορά ε, την απόρριψη των νερών στον ειρηνικό έχει αναφερθεί, χαρακτηρίστηκε από την παρέτηση του αρμοδίου υπουργού. Εμεί θα ψηφίσουμε κατά τη αντίρρηση αυτή γιατί θεωρούμε ότι οι πολίτε πρέπει να προστατεύονται από όλου του κινδύνου καρκίνου. Από αυτόν όπω και όλου του υπόλοιπου συζητήθηκαν παλιότερα Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τεράστιο σχέδιο καταπολέμηση του καρκίνου και εδώ στο Κοινοβούλιο και να αφήνουμε τον κίνδυνο τη ραδιενέργεια. Όπω είπατε, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη κατανόηση. Οπότε θα υποστηρίξουμε, υπέρ, θα υποστηρίξουμε αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστούμε για το ID. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ προσωπικά και πολύ μάλλον στην ομάδα μου ε, δεν είναι υπέρ των διακρίσεων να υπάρχει δηλαδή ένας πολιτικός σεχταρισμό. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την αντίρρηση, κυρία Ριβάζη, θα την υποστηρίξουμε, διότι η υγεία ε, πάει πέρα από την πολιτική και τα στοιχεία που μα έδωσε η κυρία Ριβάζη, αλλά και η θεμητή υποψία, ε, αυτός είναι ο όρος, έτσι, ε, συχνά έχουμε συζητήσει επικειμένων ε, όπου οι μελέτες δεν υποστηρίζουν τα επιχειρήματα και η αρχή της προφύλαξης ε, σχεδόν, σχεδόν συνεχώς παρακάμπτεται. Όταν μιλάμε όμως για κίνδυνο, για καρκίνο, και δεν μπορεί να πει το αντίθετο ο συνάδελφος, βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο ενός κινδύνου με πολυπαραγοντικού. Ο κάθε κίνδυνος λοιπόν συσσωρευόμενος μαζί με του άλλους κινδύνους μας κάνει να είμαστε πιο απαιτητικοί, πρέπει να είμαστε απαιτητικοί ακόμα και αν τα στοιχεία είναι κάπως καθυσυχαστικά. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστώ για το ECR. Ε, we disagree with the objections. Διαφωνούμε με την ε, αντίρρηση καθώς θεωρούμε ότι είναι αυθαίρετες οι επιλογές καθώς από την άλλη θεωρούμε ότι οι Ιαπωνικές αρχές εφαρμόζουν πολύ αυστηρά κριτήρια ελέγχου, πιο αυστηρά από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης ότι δεν έχει βρεθεί μη συμμόρφωση κατά τους ελέγχους εδώ και πάνω από 7 χρόνια. Ευχαριστούμε για τον Κούε. Eh, Ευχαριστώ. Ε, Ξέρουμε όλοι τα τρόφιμα που παράγονται γύρω από τη Φουρκουσίμα ε, ότι τα ψάρια της περιοχής ε, ε, δεν ελέγχονται παρκώς για την ραδιενέργεια, παρά τις διάφορες δημοσιεύσεις για την διατροφή. Και βασιζόμαστε εδώ σε αυτά που λένε οι αρχές της Ιαπωνίας και όχι στις δικά μας δεδομένα. Μπορεί η Κομισιόν να μας επιβεβαιώσει ότι τα τεστ δεν καλύπτουν το σύνολο της ε, ραδιενέργειας και της ακτινοβολίας. Ένα ε, ε, πολύ μεγάλο ποσό, μεγάλες ποσότητες ε, νερού ψήξης θα απελευθερωθεί και αυτό είναι επικίνδυνο και για διατροφική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν διευκρινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει η Ιαπωνία να αλλάξει άποψη σε ό,τι αφορά αυτό το νερό το οποίο θα, διαχει, θα διαχέεται στον ωκεανό. Μήπως θα μπορούσαμε τελικά, είναι δυνατόν ε, να έχουμε ένα τόσο ε, νοσηρό ε, μηχανισμό στα πλαίσια της Συμφωνίας των Συναλλαγών, ε, μπορούμε να διακυβεύσουμε έτσι τη διατροφική ασφάλεια και την υγεία, διατροφική υγεία, πώς είναι δυνατόν πάση θυσία να θέλουμε να προωθήσουμε το εμπόριο με μια χώρα όπως η Ιαπωνία, η οποία έχει ξεκινήσει και την σεζόν της, του κυνηγιού για τις φάλαινες, έτσι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν υπέρ αυτής της αντίρρησης. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας, παρακαλώ, έχεις το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει περιοριστικά μέτρα για την εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών από την Ιαπωνία με στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών. Κάθε δύο έτη ε, επανεξετάζονται αυτά τα μέτρα γίνεται πολύ αυστηρός έλεγχος για το, για το κέσιο, ε, για το κέσιο 134 και 137 και την επίδρασή του στη γεωργική παραγωγή. Τα αποτελέσματα ραδιενέργειας των ελέγχων έχουμε πάνω από 300.000 ε, δείγματα ε, που έχουν ε, αναλυθεί από το 2011 και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεξάγουν ελέγχους σε σχέση με τη ραδιενέργεια των τροφίμων και των ζωοτροφών που προέρχονται από την Ιαπωνία και όπως σας είπα δεν έχει παρατηρηθεί μη συμμόρφωση από τον Ιούνιο του 2011 και μετά. εστιάζουμε ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα κριτήρια κατά την επανεξέταση και βασιζόμαστε στα λεπτομερή στοιχεία που μας προσφέρουν οι Ιαπωνικές αρχές. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεξάγουν ελέγχους κατά την εισαγωγή. Σε ό,τι αφορά ε, τις, ε, διάφορες, τους διάφορους δήμους, τις διάφορες περιφέρειες, προτείνουμε να επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο εφόσον δεν έχει εντοπιστεί καμία μη συμμόρφωση το τελευταίο έτος από τη συγκεκριμένη περιοχή και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή αναλυτικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την Φουκουσίμα και την περιοχή αυτή, έχουμε θέσει το όριο να μην υπάρχουν μη συμμορφώσεις τα τελευταία δύο έτη. Όπως ανέφερε και η κυρία Ριβαζή, τα μέγιστα όρια που ισχύουν για τα τρόφιμα από την Ιαπωνία είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με αυτά που εφαρμόζει και το Τσέρνομπιλ, για παράδειγμα. Ή αυτά που θα εφαρμόζονταν αν υπήρχε κάποιο πυρηνικό ατύχημα στην Ευρώπη. Οι αλλαγέ στον εκτελεστικό κανονισμό τη Επιτροπή βασίζονται σε εκατοντάδε χιλιάδες αναλυτικά αποτελέσματα σε σχέση με τη ραδιενέργεια διαφόρων τροφίμων με εξαίρεση το βόηο κρέα και σε περίπου 130.000 ε, ε, ε, δείγματα σε βόηο κρέας από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 έχει γίνει λεπτομερής ανάλυση των εν λόγω στοιχείων και τεκμηρίωση των αλλαγών και μάλιστα ε, στα, μπορούμε να σας προσφέρουμε και την απαραίτητη τεκμηρίωση εφόσον το ζητήσετε. Η Επιτροπή επαληθεύει συνεχώς τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγουν οι Ιαπωνικές αρχές καθώς και τα αποτελέσματα των ε, ελέγχων στις εισαγωγές και φυσικά ε, αφόσον προκύπτουν νέα στοιχεία αναθεωρούμε την κατάσταση. Ενημερωνόμαστε συνεχώς για την κατάσταση του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, τον Ταϊτζή, καθώς και για την χρήση του νερού ψήξης σε αυτόν τον σταθμό. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να ενημερώνουν την Επιτροπή σε σχέση με οποιαδήποτε εξέλιξη ε, σε ό,τι αφορά το αποθηκευμένο νερό ψήξης. Ανάλογα λοιπόν με τις εξελίξεις και εμείς θα δράσουμε έχει την άποψη η Επιτροπή ότι με την εφαρμογή των αυστηρών αυτών ε, κριτηρίων και με βάση τα διαθέσιμα κριτήρια ο προτινόμενος κανονισμός συνεχίζει να διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών και πιστεύουμε ότι η Επιτροπή δεν υπερβαίνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες που ε, προκύπτουν από τον κανονισμό 1078 του 2002 για την σύνταξη αυτής της πρότασης. Ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη το 9 για, τις, ε, για τα ζανιοκτώνα. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Χάζενκαμπ και μετά τη λιμέτια του πράσινου. Κυρία Χάζενκαμπ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς για άλλη μια φορά πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για τις διαδικασίες παράτασης της αδειοδότησης για διάφορα ζενιοκτώνα. Παλιότερα, μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε την αντίρρησή μας και ζήτησε να μην υπάρξουν νέες παρατάσεις για τα ζενεοκτώνα, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, για τα ζώα και για το περιβάλλον. Λίγες μέρες αργότερα, για άλλη μια φορά η Κομισιόν προέβησε σε παράταση. Μιλάμε για μια παράταση ενός έτους για διάφορες ουσίες. Η παράταση αυτή υποτίθεται ότι είναι απαραίτητη διότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αλλά γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με τις ε, Ολλανδικές αρχές, για το Μαγκοζέπ υπάρχουν αρκετά δεδομένα στην ΕΦΣΑ για να λυθεί απόφαση τώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικά πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξης ε, αδειοδότησης τέλη Ιανουαρίου, διότι το ΜΑΚΟΣΕΠ είναι το ζενευτόν που χρησιμοποιείται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί πολλές ασθένειες στις κατοχώρες και στη Γαλλία, όπου χρησιμοποιήθηκε ευρέω από τους γεωργού. Υπάρχουν σοβαρέ ενδείξεις που δείχνουν ότι οι γεωργοί και οι οικογένειές τους ε, υποφέρουν πολύ συχνότερα από ασθένειες, από νόσους Πάρκινσον, από τι αλλού. Ε, δεν λέμε όχι μόνο για νευροτοξικές ασθένειες, αλλά διαπιστώθηκε ότι δημιουργεί πρόβλημα και στην αναπαραγωγή δεν πλήρει λοιπόν ε, τα κριτήρια ασφαλείας ε, που προβλέπονται στον κανονισμό για τα ζανιοκτών. Αυτό η τοξική ουσία θα πρέπει να απαγορευτεί το συντομότερο δυνατόν και είναι απολύτω ανεύθυνο να εκθέτουμε ακόμα για άλλο ένα χρόνο του ανθρώπου σε αυτή την ε, δραστική ουσία. Το ίδιο ισχύει και για το ντεξτροστρομίν. Στον κανονισμό του 2015 διαπιστώνουμε ότι δημιουργεί ορμονικά προβλήματα τέτοιου είδου ουσίε ε, δεν πρέπει να λαμβάνουν παράταση. Αυτό αντίκειται για άλλη μια φορά στην ε, νομοθεσία για τα ζυζανιοκτώνα. Η Κομισιόν πρέπει οπωσδήποτε αυτό το μήνα να ξανακάνει ε, προτάσει απαγόρευση αυτών των επικίνδυνων ουσιών. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα αφού υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που αιτιολογούν τέτοια απαγόρευση. Αλλά επίση και διότι η Κομισιόν με αυτέ τι διαδικασίε για άλλε ουσίε μπορεί να δείξει ότι ε, μπορεί και να το κάνει. Οπότε αναμένω την απάντηση της Κομισιόν για αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε για το ΕΛΚ. Αγαπητέ Πρόεδρε, καταλαβαίνω ε, τους λόγους. Ε, πρόκειται για καρκινογόνες ουσίες, ε, οι οποίες πρέπει να περιοριστούν και τοξικές ουσίες. Η παράταση των αδειών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες. Επιστημονικά στοιχεία φυσικά Ωστόσο, αυτό, η πρόταση εδώ αφορά την παράταση τη ασυδότησης για 10 ουσίε που αυτή τη στιγμή έχουν άδεια. Η αξιολόγηση και η έλεγχη και οι σχετικέ διαδικασίε δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε κάποια απόφαση. Η νομική κατάσταση σε αυτέ τι περιπτώσει είναι σαφή. Η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να ανανεώσει την αδειοδότηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που εξετάζει η παραγωγή αυτών των προϊόντων αυτή η παράταση θα γίνει αφού γίνει η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ. Η απόφαση για την αδειοδότηση θα διαρκέσει τους μήνες που θα διαρκέσει μέχρι να ληφθεί η απόφαση της ΕΦΣΑ. Η υποστήριξη σε αυτό το ψήφισμα ε, θα σημαίνει ότι θα απογορεύσουμε την κυκλοφορία χωρίς να υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση θα λέμε ότι αυτέ οι ουσίε δεν μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά ε, διαλύματα που χρησιμοποιούν οι γεωργοί πολύ αποτελεσματικά για τι επιχειρήσεις του. Ένα τέτοιο βήμα θα οδηγήσει επίση στο ότι πολλοί γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με Γεωργού τρίτων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία παράγει με πολύ αυστηρά πρότυπα τα καλύτερα τρόφιμα. Οπότε αυτό το ψήφισμα θέτει σε κίνδυνο τους γεωργού μας και την ασφάλεια σχεδιασμού και της γεωργίας. Οπότε εγώ λέω να απορρίψουμε αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστέ. Παρακαλώ. Όχι. Για το Renew. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ Έχουμε ζυζανιοκτώνα με, άλλα, με άλλες ουσίες που είναι προβληματικές, αλλά άλλες είναι και άλλες δεν είναι και τα έχουμε, έχουμε βάλει μαζί. Το Μακοζέπ, παραδείγματος χάρη, αλλά και μια άλλη που δεν μπορώ να προφέρω καλά, τη Μοξιστροβίν. Ε, ξέρουμε ότι αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια για την αδειοδότηση. Αφενός λοιπόν υπάρχει μια πίεση να παραμείνουν στην αγορά όσο γίνεται περισσότερο ε, τραβώντας την αξιολόγηση, παρατείνοντάς της. Ε, η Κομισιόν από την άλλη θα πρέπει να ακολουθήσει την οδό που έχει ακολουθήσει πολύ σωστά για, άλλα, για άλλες ουσίες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για δύο ουσίες που είναι προβληματικές εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντικατασταθούν αυτά τα επικίνδυνα ζωνιοκτώνα. Για την ID δεν θέλει κάποιο το λόγο, για την ECR. Ναι, εμεί είμαστε κατά τη αντίρρηση. Η προβλεψιμότητα για τους γεωργούς ε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Μιλάμε απλά λοιπόν εδώ για μια παράταση που δίνεται και δεν καταλαβαίνω που δράζει αυτή η αντίρρηση για τους πράσινους. Α, ωραία, θα κλείσω εγώ. Ε, ε ακούστε, θα είμαι σύντομη. Μου κάνει εντύπωση που έλεγχαν κάποια πράγματα. Το μανκουζέπ και το ντιμοξιστρομπίν πάντως είναι ενεργές ουσίες που υπάρχουν στα ζανιοκτώνα. Είναι γνωστό ότι έχουν τοξικά ε, χαρακτηριστικά, ότι είναι ενδοκρινικοί διαταρακτές ε, έχουν κατηγοροποιηθεί ως, ε, ε, ως τέτοιες. Παρ' όλα αυτά αδειοδοτούνται χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτιολόγηση παραβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σύμφωνα με την νομοθεσία όλες οι ουσίες ετροτοξικές δεν πρέπει να επιτρέπονται και θα πρέπει να περιορίζονται χρονικά οι όποιες άδειε. Εφόσον υπάρχουν δηλαδή αποδεικμένοι κινδυνικοί για την υγεία και για το περιβάλλον, η ανανέωση αυτών των δύο ουσιών τρεις φορές ήδη ε, μας δείχνει ότι η Κομισιόν δεν βάζει την υγεία και την ε, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας πριν από τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει αυτή την παράταση, τουλάχιστον για αυτές τις δύο ουσίες. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία τη Υγεία παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλό απόγευμα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, ε, να πω ότι κατά την άποψή μας δεν έχουμε ξεπεράσει τις εξουσίες της Εφαρμοστικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτό το μέτρο. Το μέτρο έρχεται με, μετά από μια διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό για τη φυτοπροστασία. Άρθρο 17, η σχετική διαδικασία, που απαιτεί όταν η έγκριση μιας ουσίας ε, είναι κοντά στην λήξη άδεια, ε, ε, τότε η Κομισιόν πρέπει να παρατείνει την έγκριση, εφόσον μας το ζητήσει ο παρασκευαστής. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής πρόσφατα, σε μια σχετική υπόθεση, επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν έχει αυτή την υποχρέωση. Και αυτό ισχύει και για τις δέκα αυτές ουσίες που υπάρχουν σε αυτό το σχέδιο κειμένου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτό το μέτρο και η διαδικασία του άρθρου 17 εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ταξινόμηση των ουσιών. Εφαρμόζεται δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις. Είτε η ουσία αυτή πληρεί τα κριτήρια, είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι η ταξινόμηση δεν δίνει σε μας επιχειρήματα ή λόγους για να μην παρατείνουμε την περίοδο έγκρισης. Δυστυχώς υπάρχουν καθυστερήσεις στη διαδικασία. Συμβαίνουν αυτά, έχουν συμβεί στο παρελθόν και αυτό βεβαίως ε, οφείλεται σε πολλούς λόγους. Συχνά έχουμε καθυστερήσεις κατά την αξιολόγηση από το κράτος μέλος. Στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Είχαμε μια παράλληλη αξιολόγηση ε, σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση του κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί όλο και πιο συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει ασυνέπεια. Είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει πλέον κάποια συνέπεια σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση με βάση την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών και που αποτελεί και βάση για τα συμπεράσματα τη ΕΦΣΑ στη συνέχεια. Αυτό όμω εξηγεί και τι καθυστερήσει στην προηγούμενη περίπτωση. Επίση, χρειάστηκαν κάποια περαιτέρω στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα με βάση την εφαρμογή των νέων κριτηρίων ε, για τους ενδοκρινικούς διαταρακτές που έπρεπε να συλλεχθούν τα στοιχεία αυτά και να αξιολογηθούν. Ε, στην, διαδικασία, στην νομοθεσία μας, όταν χορηγηθεί έγκριση ή ανανέωση, πρέπει να πληρεί τα κριτήρια. Πρέπει να είναι ασφαλές για τον καταναλωτή, για το περιβάλλον, για τα ζώα. Θα γίνει μια σε βάθος αξιολόγηση για αυτά τα δύο προϊόντα τα οποία υπάρχει ανησυχία, το Μανκοζέπ και το και η Δημοξιστρομπίνη. Για το Μανκοζέμπ έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ. Έχουμε τα συμπέρασματα της ΕΦΣΑ που ολοκληρώθηκαν. Η αξιολόγηση κινδύνου δεν έχει πάρθει ακόμα σχετική απόφαση. Θα γίνει και αυτό το συντομότερο δυνατόν. Τώρα για την Δημοξιστρομπίν ε, ακόμα υπάρχουν κάποια στοιχεία για τους ανδοκρινικού διαταρακτέ και τις σχετικές ε, ιδιότητες που είναι προς αξιολόγηση. Αυτό είναι προς όφελο των καταναλωτών ε, θα βοηθήσει τον καταναλωτή, θα βοηθήσει την ΕΦΣΑ να πάρει μια ε, στοιχειοθετημένη απόφαση. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι κάποιες περαιτέρω πληροφορίε ε, και κάποιε παράλληλε διαδικασίε οδήγησαν σε καθυστερήσει. Το σημειώνουμε αυτό, αλλά για την προστασία τη υγεία των καταναλωτών είναι σημαντικό όλε οι θέσει πληροφορίε ε, να μπορέσουν να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή ποια απόφαση θα πάρθει σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου για αυτέ τι δύο περιπτώσει. Θέλω πάντω να σα ε, διασφαλίσω ότι όποια απόφαση που θα έρθει θα, θα βασιστεί σε επιστημονικά δεδομένα και σε ένα πνεύμα προστασία του καταναλωτή, ε, του περιβάλλοντο ε, και των ζώων. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Ξεκινούμε 9.30 αύριο το πρωί με την επικεφαλής της EIB, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στη συνεδρία των συντονιστών.